Good afternoon, ladies. κυρίες και κύριοι. Καλώς όρισατε αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να αρχίζουμε σιγά σιγά τη σημερινή μας συνεδρία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρώτο θέμα έγκριση ημερήσιας διάταξης. Έχετε προτάσεις, υποδείξεις, επιθυμίες για αλλαγή της ημερήσιας διάταξης. Όχι. Από ό,τι βλέπω και σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Επόμενο θέμα, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 11 έως 14 Ιανουαρίου, καθώς επίσης και της 25ης. Κοινή συνεδρίαση που κάναμε με την Επιτροπή ΚΟΤΕ στις 25 Ιανουαρίου. έχουν διανεμηθεί, μάλλον και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο ε, τα πρακτικά. Ε, η συνήθιση διαδικασία ισχύει αν δεν εκφραστούν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίας θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Ούτε προτάσεις, ούτε σχόλια, ανακοινώσεις Προέδρου καμία, δεν έχω καμία ειδική ανακοίνωση να σας κάνω σήμερα, οπότε και θα προχωρήσουμε όπως είμαστε εις το επόμενο θέμα. Επανεξέταση του ρόλου του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Είναι το πρώτο ουσιαστικό θέμα μας ε, για σήμερα. Μελέτη που θα παρουσιαστεί από τον καθηγητή Τζον Μπάχτλερ για την ε, πολιτική συνοχής. Η Επιτροπή μας ανέθεσε αυτή τη μελέτη λοιπόν το κέντρο ερευνών μαζί με το Πανεπιστήμιο του Στραθκλετ. Στόχος είναι να έχουμε μια συνολική ανάλυση και αξιολόγηση για το πώς οι στόχοι της περιφερειακής πολιτικής έχουν επιτευχθεί με μέσα ε, στα οποία συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η μελέτη θεωρεί ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην πολιτική συνοχή έχει αυξηθεί σημαντικά στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 και συνέχισε να αυξάνεται στη νέα προγραμματική περίοδο. Επίσης καταλήγει η μελέτη ότι είναι παρεξηγημένη η συνεισφορά της στην πολιτική συνοχής. Και προτείνει ότι για να αυξηθεί η λογοδοσία και η διοργανική σχέση με την Επιτροπή μας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να συσφίξουμε τους δεσμούς. Έχουν έρθει να μας παρουσιάσουν τη μελέτη δύο από τους ε, ηθήνοντες που την ανέλαβαν, ο καθηγητής Τζον Μπάχλερ και ο κύριος Άρνο Βαντερσφέτς και οι δύο του Πανεπιστημίου του Strathclyde. Strathclyde. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στους δύο προσκεκλημένους για τη σύντομη παρουσίαση από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde και οι δύο μαζί 30 λεπτά ή 10-15 έκαστος έτσι και μετά συζήτηση και ερωτήσεις. Who of you will begin. Ποιο θέλει να αρχίσει από εσά, παρακαλώ. Ο κύριος Μπάχτλε. Um, Στο Πρόεδρε, μέλη τη Επιτροπής, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Uh, για να μα παρουσιάσουμε τη μελέτη, είμαι ο Τζον Μπάχτλερ και ξεβονίμων ο δόκτων Άρνο Βαντεσβέτ, ο οποίο ηγήθηκε τη μελέτη που θα παρουσιάσουμε, αναθερώντας το ρόλο Τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του σχετικού ομίλου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτική συνοχή. Ποιο είναι το πλαίσιο της μελέτης που τα ανέφερε και η πρόεδρος ο Ο αυξανόμενος ρόλος της Ευρωπαϊκής τάπες Επενδύσεων στην πολιτική συνοχής, άμεσα και έμεσα με ένα ευρυνόμενο φάσμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Συνεπάγεται αυτό δανειοδότηση, δημιουργία δυναμικού, συμβουλές, αναλυτικές υπηρεσίες και εφαρμογή χρηματοπιστωτικών ε, μέσων, χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων. Και αυξάνεται ο ρόλος αυτός. Και αυτό οδηγεί σε ερωτήσεις που αποτελούν και βάση των μελετών μας. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται καλύτερη κατανόηση τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Και εξ αυτού το ερώτημα το εξή. Αυτή η δραστηριότητα είναι αποτελεσματική, τουλάχιστον όσο την εκτιμούμε σχετικά με την πολιτική συνοχής. Μετά, ποια είναι η λογοδοσία, ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, πόσο διαφανής, πόσο ορατές οι δραστηριότητες της και οι υπηρεσίες της και υπάρχουν και διοργανικά ζητήματα σημαντικά. Σχέση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σχέση Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Επενδύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνάρτηση με την πολιτική συνοχή. Και απορρέει και το εξή ερώτημα. Ποιε είναι οι συνέπειε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πολιτική συνοχής και όσον αφορά την Επιτροπή σας πιο συγκεκριμένα. Στόχος της μελέτης ήταν αυτά τα ερωτήματα και οδηγήσαν στη δομή της παρουσιάσεως που θα δείτε. Προσέξτε το εξής. Η μελέτη είναι απλό σχέδιο τελικής εκθέσεως. Χρειάζεται περαιτέρω χτένισμα το κείμενο. Λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα σχόλια άλλων θεσμικών οργάνων και σχόλια και πληροφορίες της Επιτροπής σας. Και θα φτάσει στην οριστική μορφή η έκθεσή της το ταχύτερο δυνατόν μετά την συνεδρίασή μας αυτή. Θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο. Αυτός θα παρουσιάσει και την ουσία της μελέτης αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη για την πρόσκλησή τους και τη δυνατότητα να παρουσιάσω τη μελέτη εδώ σήμερα. Ξεκινώ λέγοντας λίγα λόγια για τη μεθοδολογία. Αφετηρία της μελέτης ήταν συστηματική αναθεώρηση των βασικών διαφόρων κειμένων που υπάρχουν σε πολιτικό πανεπιστημιακό επίπεδο. Ανάλυση δηλαδή των διαφόρων χρηματοστικών μέσων και των πρωτοβουλειών στην πολιτική συνοχή στην περίοδο 2007-2013. Εκεί έπαιξε ρόλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λαμβάνοντα υπόψη τα στοιχεία τη συνοπτική εκθέσεω για τα χρηματοστικά μέσα. Άλλο στοιχείο που λάβαμε υπόψη. Κάναμε σύγκριση χωρών σε επαφή με ανώτου εξωματούχου που ήταν υπεύθυνοι για την πολιτική συνοχή. Αναλύσαμε 28 κράτη-μέλη. Πήραμε 19 απαντήσει από τα κράτη-μέλη. Θέλαμε να αναλύσουμε τι διοργανικέ σχέσει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω συνεντεύξεων και επαφών με κροσόπου των φορέων αυτών. Συναθρήσαμε τι πληροφορίε. Καταλήξαμε στη συνοπτική έκθεση. Και έχουμε συστάσεις και συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Στρέφουμε τώρα προς το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην πολιτική συνοχής έχουμε χωρίσει τις δραστηριότητε σε κατηγορίες, σε τέσσερις κατηγορίες. Υπάρχει και κάποια επικάλυψη μεταξύ κατηγοριών. Δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ κατηγοριών. Πρώτα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από την αρχή τη πολιτική συνοχή δανειοδοτούσε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω τη πολιτική συνοχή. Η τράπεζα προσφέρει διάφορα είδη δανείων. που τα βλέπετε στην έκθεση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, άμεσες δανειοδοτήσει, ενδιάμεσες δάνεια πλαισίου και έχουμε και υποσύστημα των διαφόρων δανείων για διαφθορτικά προγράμματα. Τα SBLs όπως αποκαλούνται. Αφορούν συγχρηματοδότηση πολλαπλών έργων και επενδύσεων που συμπεριλαμβάνονται σε επιχειρησιακά προγράμματα και τα διαφθορτικά ταμεία. Δεύτερη κατηγορία είναι η δημιουργία δυναμικού σε κάποιες περιπτώσεις η δανειοδότηση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εξαρτάται από απαιτήσει για τεχνική αρρωγή. Να υπάρχουν μονάδες εφαρμογής έργου, υλοποίησης έργου Φερρυπίν. Και στα πλαίσια των πολιτικών συνοχής, το Jaspers θεσπίστηκε το 2005, κοινή πρωτοβουλία της DG Regio και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το Jasper είναι κοινή βοήθεια για υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και δημιουργούν το ακρόνιμο Jasper. Το Jaspers δίνει συμβουλές ανεξάρτητες σε 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τρεις χώρες IPA για να γίνει σύγκριση των έργων ποιότητας. Η πρωτοβουλία Jasmine ήταν άλλη μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε το 2007 για να βοηθήσει μικροχρηματοδοτικούς οργανισμούς που δεν είναι τράπεζες να αυξήσουν την κλίμακα των αστηριοτήτων για να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα όσον αφορά τα έργα μέσα μικροχρηματοδοτήσεως. Και για την περίοδο 2014-2020 έχουμε μια νέα βάση για τεχνική αρρωγή που θα δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σύμπραξη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τα χρηματοδοτικά μέσα που καλύπτουν όλη την υλοποίηση, όλο τον κύκλο εφαρμογή των μέσων αυτών. Τρίτος ρόλος της τράπεζας. Παρέχει συμβουλές και αναλυτικές υπηρεσίες όσον αφορά τα προγράμματα, τις αρχέ για την εφαρμογή πολιτικών συνοχή. Και επεκτάθη ο ρόλος αυτός ε, όταν διαδεχόταν τα προγράμματα το ένα το άλλο και είμαστε στο πλαίσιο της ειδικη υποστηριξης υποστήριξης 2007-2013, προγραμματική περίοδος αυτής, και το EIF έκανε ανάλυση για τα ε, διάφορα μέσα επιχειρήσει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έκανε μελέτες, εφικτο, το, μέσω των πρωτοβουλίων Τζέσικα και 2014-2020 είναι υποχρεωτικέ εκ των υστέρων να λύσει τεχνομετωστικά μέσα που έχουν στηρίξει από τα εθνικά προγράμματα και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ανέπτυξε τη μεθοδολογία για τι εκ των υστέρων αναλύσει και μπορεί, αν ζητηθεί από τι διοικητικέ διαχειριστικέ αρχέ, να γίνει υπεύθυνη για την διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να εφαρμόζει ε, να διαθέτει αυτούς τους πόρους για τα μέσα αυτά τα χρηματοστικά. Κάτι που προλέπεται από κάτι μέλη και τις περιφέρειες. Όταν γίνει αίτηση από τις περιφέρειες και τα κάτι μέλη, είναι υποχρεωτική διαχείριση, εντολή για διαχείριση μάλλον. Για αστική ανάπτυξη και για άλλα έργα. Και για την περίοδο 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παίζει ρόλο για την εφαρμογή μέσων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την πολιτική συνοχή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως η πρωτοβουλία της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Τώρα στρέφουμε τώρα προς τα χρηματοστικά αυτά μέσα. Η μελέτη ελέγχει τις ευρύτερες δραστηριότητες τη Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά εστιάζεται όλους ιδιαίτερο στα χρηματοστικά μέσα και πολύ σύντομα τα μέσα αυτά είναι μέτρα ε, οικονομικής υποστηρίξεως που πιστεύονται αυτά τα χρώματα μπορεί να είναι αξιόγραφα που δίδονται, δάνεια, εγγυήσει, διάφορα μέσα επιμερισμού του κινδύνου και μπορούν να συνδεθούν, να συνδυαστούν και με χορηγίες ε, και δωρεές ε, άμεσα μπορεί να υπάρχει αυτή η επαφή ή μέσω και διαφόρων ταμείων που δημιουργούνται με στόχο τη συνεισφορά και την υποστήριξη σε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Και βλέπετε από τις διαφάνειες. Στην πολιτική συνοχής έχει αυξηθεί η σημασία των χρηματοστικών μέσων αυξήθηκε από 570 εκατομμύρια από την 94-99 την περίοδο αυτή και πήγε στα 1,3 δις την περίοδο 2000-2006, 2007-2013 πήγε στα 17 δις και η αναλήψη υποχρεώσεων για την περίοδο 2014-2020 είναι περίπου στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα η αυξανόμενη χρήση αυτών των μέσων οδήγησε σε πιο συγκεκριμένη ένταξη, συμπερίληψη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της χρηματοστικής ενισχύσεως. Έχει από τη μεταρρύθμιση ιδιωτικών ταμείων έχει συμμετάσχει στην ενοποίηση των έργων αυτών. Πριν το 2000 δεν υπήρχαν διατάξει συγκεκριμένε για να, να συμπεριλαμβάνεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεω στην υλοποίηση των διαρθωτικών ταμείων. Εθεωρείται σαν ένα πάροχο χρηματοστική βοηθεία μαζί με τα ιδιωτικά ταμεία. Ε, το 2006 ήταν παρόμοιο ο ρόλο, περίοδο 2006, δόθηκε εντολή όμω για την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσία, άρα έπρεπε να συμμετέχει σε επιτροπέ, εποπτεία και ε, συμβούλευε στην προετοιμασία των διαφόρων ε, εγγράφων προς τα προγράμματα. Έπαιξε πιο ουσιαστικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην υλοποίηση και την χρήση των χρησιμοποιητικών μέσων την περίοδο 2007-2013, πιο συγκεκριμένα στον αφορά τη διαχείριση. Ήταν ένα νέο ρόλο που συνετέθη στα πλαίσια τη πολιτική συνοχή και στην αρχή του την αρχή της περίοδου 2017-2013 μνημόνια επεγράφησαν όσον αφορά το Τζέσικα και το Τζάσπερ και λοιπά που υπεγράφησαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τάξη Επενδύσεων και άλλου ευρωπαϊκού Στην περίοδο 2014-2020 του κανονισμός προβλέπει επίσης το ρόλο της Ευρωπαϊκής τάπες Επενδύσεων για τη χρήση των μεσών και διαφόρων άλλων μέσων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως έχει συμβουλευτικό ρόλο για τα διάφορα προγράμματα και ο ρόλος αυτός καθορίζεται σαφώς στον κανονισμό. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο ότι παρόλο που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αυξημένε ε, ευθύνε όσον αφορά την υλοποίηση και την χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στην πολιτική συνοχή, για τη διαχείριση των διευθυντικών ε, ταμείων, αυτή είναι ευθύνη του κράτου μέλου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την κοινή διαχείριση, όπω αποκαλείται. Τώρα πάμε τώρα στην αποτελεσματικότητα του συμβουλευτικού ρόλου τη Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων, η δημιουργία δυναμικού. Κάναμε αναλύσει όσον αφορά τι ελλείψει που υπάρχουν. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το, στα πλαίσια του Τζέρεμι και του Τζέσικα έκαναν αναλύσει και οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορεί εκτίμησαν τι προσπάθειε. Η ανάλυση μα δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έκαναν μελέτε και συστάσεις που όμως ε, δεν συμμορφωνόταν οι αρχές οι εθνικές και οι τοπικές με αυτές τις ε, συμβουλές. Και δεν ξέρουν πόσο αποτελεσματικές ήταν οι μελέτες γιατί ήταν και πολύ δαπανηρές. Όμως ε, οι μελέτες εθεωρήθησαν ότι ήταν σημαντικό βήμα προωθώντας την χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και μπορεί να θεωρηθεί σε ένα πρώτο βήμα προς το, προς το να κινητοποιηθούν οι αρχές διαχείρισης και τα κράτη-μέλη και να δουν πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα εργαλεία και να δημιουργήσουν μια συνένεση γύρω από την προσέγγιση της χρήσης των μέσων αυτών. Και κάτι άλλο που ανέφερα είναι πώς φαίνονται, γίνονται τελειπτά ε, τα, οι συγκρούσεις συμφερόντων στον αφορά της εξολογής Ευρωπαϊκής Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων όσον αφορά τις μελέτες σκοπιμότητας και της αξιολογήσεως και όσον αφορά τη διαχείριση των ταμείων. Αυτό μπορεί να ιδωθεί στο εξή πλήσιο Ότι οι πρωτοβουλίε Τζέρεμι και Τζέσικα ήταν πιλωτικέ πρωτοβουλίε και οι δομέ ε, ήταν ε, εξελισσόμενε και σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να αναφέρουμε στο τέλο η διαχειριστική αρχή του κράτου μέλου αποφάσισε επί ε, τη όλη δομή και τη διάθρωση τη χρήσεω των πόρων και ποιο θα είναι διαχειριστή των πόρων. Και τέλο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανταποκρίθηκε σε κάποιε απαιτήσει του διπλού ρόλου που είχε, αναθέτοντα διαδικασίε αξιολόγηση, αλλά με κεντρική ανάληψη ευθυνών για την εκ ανάλυση για την περίοδο μέχρι το 2014. Τώρα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, όσον αφορά τη διαχείριση της εντολής που της ανετέθη. Τώρα, αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και όσον αφορά το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων είναι κάτι ε, πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο γιατί δεν είχαμε πάρα πολλά στοιχεία. Είχαμε και σύντομο χρονικό διάστημα για την ανάλυση και μικρή εμπειρία όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των χρηματοστικών μέσων. Βασιστήκαμε εμεί στα στοιχεία που μα δώσαν τα κράτη-μέλη στι συνοπτικέ εκθέσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω και για τα έτη 2000, το 2014 είδαμε ότι είχαμε χαμηλότερα επίπεδα απορρόφησης βλέποντας την απορρόφηση των πόρων από τους τελικούς αποδέκτες εν συγκρίση με ε, τα ταμεία που δεν είχαν σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ίσως ο ρυθμός απορρόφησης που ήταν περιορισμένος να οφείλεται στο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι αμεμειγμένη με κράτη-μέλη που έχουν μικρότερες δυνατότητες ή ε, που είχαν πληγεί όλος ιδιαίτερος από τη χρηματοστατική κρίση και αυτό οδήγησε καθυστερήσει σε άλλη εξήγηση. Το νομικό πλαίσιο για τα χρηματοστατικά μέσα για το 2007 μέχρι το 2013 ε, δημιούργησε διάφορα προβλήματα σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έτσι, δεν περαιτέρω σημειώνεται ότι ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ο τρόπος, ο εσωτερικός έλεγχος των φορέων αυτών δείχνει πολύ ψηλότερο επίπεδο για την περίοδο 2015 όπου βλέπουμε μια ε, ακμή αν θέλετε στο γράφημα για τις απορρόφησεις Άλλο θέμα ήταν ε, τα τέλη διαχείρισης και από τα στοιχεία που έχουν τη Συνοπτική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε ότι ε, το κόστος διαχείρισης για, αντιστοιχούν με τους θεσμούς που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν συγκρίνουμε τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με φορείς εκτός αυτών, βλέπουμε ότι τα τέλη διαχείριση το κόστος διαχείρισης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ψηλότερο. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και των άλλων φορέων εκτός αυτού και αυτό εξηγείται διότι υπάρχουν διαφορετικά τέλη και διαφορετικό κόστος διάφορα προϊόντα για τα διάφορα αξιόγραφα είναι πιο ψηλό το κόστος από εκείνα που είναι για εγγυήσεις και δανειοδοτήσει. Και υπάρχουν ιδιαιτερότητε που αφορούν τα ταμεία και τι χώρε και διαφορέ ίσω να καθορίζουν την τελική δομή του κόστου διαχείριση. Τώρα, όσον αφορά τη δανειοδότηση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, ε, επηρεάζει πολύ τι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή ε, Ενώσεω και ο αντίκτυπο έχει αυξηθεί τι τελευταίε δεκαετίε τώρα στην παρούσα μορφή παίζει διπλό ρόλο. Πρώτα απ' όλα έχει πρόσβαση, είναι σαν επενδυτική τράπεζα που πρέπει να είναι, να έχει, να είναι αξιόπιστη και να έχει βαθμολόγηση τριπλού α και μπορεί να δίνει δάνεια σε χαμηλότερο κόστος στους δανειστές. Μετά είναι δημόσιο θεσμικό όργανο και θα πρέπει να υλοποιεί ευρύτερου στόχου πολιτική Ευρωπαϊκή Ενώση. Οι δανειοδοτικέ τη δραστηριότητε αντικατοπτρίζουν το διτό τη ρόλο Τώρα για το 2007-2013 ε, η συνολική συνεισφορά στην, στους στόχους οικονομικής και κοινωνικής συνοχής ήταν 147 δισεκατομμύρια. Βλέπετε από κάτω τους βασικούς αποδέκτες, ποιες είναι οι χώρες που δέχτηκαν αυτά τα ποσά δανειοδοτήσεως. Η κλίμακα της χρηματοδοτήσεως δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παράγει, οικονομικά ε, προϊόντα που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ενώσης και τις δαπάνες. Όμως υπάρχουν Κάποιε μελέτε ανεξάρτητε πανεπιστημιακέ όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχει εδώ τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κυρίω σε σχέση με την πολιτική συνοχή, η κλίμακα τη ανδιοδοτήσεω για έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω πολιτική συνοχή δεν είναι κάτι εύκολα αντιληπτό. Δεν υπάρχουν ομαδοποιημένα στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω που να δίνουν μια γενική εικόνα τη χρηματοδοτήσεω για την πολιτική συνοχή και τα σχετικά έργα. Ανοίξουμε τώρα μία ματιά στις ε, απαντήσεις από τα κράτη μέλη Και αυτό το οποίο κάνει το Ταμείο αλλά και η Τράπεζα είναι να <clears throat> προσπαθούν να ικανοποιήσουν ε, τι επιδόσει των μελών. Πρώτα πρώτα όσον αφορά τη δημιουργία δυναμικού και όσον αφορά συμβουλευτικέ ε, υπηρεσίε και πάμε περίπου στο 4 με άριστα το 5. Επίσης έχουμε και το θέμα της διαχείρισης των ε, πόρων και των ταμείων, οπότε βλέπουμε ότι εκεί πέρα οι επιδόσεις, η βαθμολογία τόσο είναι λίγο πιο χαμηλή αυτή η διαφάνεια είναι λίγο πιο μικρή, αλλά τέλος πάντων οι ερωτώμενοι πρέπει εδώ να βυσμάνουν σε ποιους ε, τομείς ε, ωφελήθηκαν περισσότερες δραστηριότητες της, της ε, τράπεζας και των προϊόντων και εδώ βλέπετε το σύνολο των απαντήσεων και το, στο που οδήγησαν βλέπουμε ότι το, τα πιο βασικά ζητήματα εδώ ήταν η προσβασιμότητα στην συγχρηματοδότηση και στην αναλυτική υποστήριξη της τράπεζας που ήταν ε, το όφελος που οι περισσότεροι ανέφεραν όσον αφορά ε, την πολιτική συνοχή. Ε, Παρομοίω έπρεπε να πούνε οι ερωτώμενοι ποιε είναι οι βασικέ ε, προκλήσει και εδώ αναφέρθηκε ως πρόβλημα βασικό η πολυπλοκότητα των κανόνων των και των κανονισμών και επ' αυτού είπαμε ότι θα πρέπει η τράπεζα να λειτουργήσει στα πλαίσια των όσων ορίζουν οι κανονισμοί και ότι βέβαια δεν φταίει η EIB, η τράπεζα, για το πόσο πολύπλοκη είναι η νομοθεσία. Όμως από την άλλη μεριά αυτό διαμορφώνει την εικόνα στα κράτη-μέλη. Επίσης είπαμε ότι είναι υψηλό το κόστος διαχείρισης αλλά και υλοποίηση εφαρμογής και αυτά είναι σημαντικά ε, προβλήματα. Of the EIB cohesion policy. Τώρα βλέπουμε τι άλλο γίνεται με την πολιτική συνοχή. Βλέπουμε ότι είναι έντονο ο τεχνικό, τεχνολογικό χαρακτήρα, ο οποίο οδήγησε σε κάποια πάρα πολύ σημαντικά ερωτηματικά όσον αφορά την, ε, ε, την διαφάνεια, όσον αφορά την προβολή των δραστηριοτήτων, αλλά ε, και τη λογοδοσία είπαμε ότι είναι αρκετά αυτόνομη η τράπεζα αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει αυτονομία θεσμικού χαρακτήρα για την IB αυτό βέβαια δεν σημαίνει όμως ότι δρά ανεξάρτητα και υπεράνω του κοινοτικού δικαίου τα τελευταία χρόνια επίσης είναι συνεχής προσπάθεια της τράπεζας να βελτιωθεί η διαφάνεια και επίσης ε, να εφαρμόσει τις συμμετοχικές αρχές ας πούμε όσον αφορά κάποιες εκθέσεις για σημαντικά διζητήματα. Εδώ έχουμε το θέμα της κοινοτομίας. Αυτό έχει βελτιώσει την ε, διαφάνεια. Παρ' όλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να αναβαθμιστούν κάποια στοιχεία της πολιτικής διαφάνειας της ε, τράπεζας, ιδίως όσον αφορά το πώς θα, αξιολογηθεί ε, η επίπτωση των δανείων. Πάντως τα κράτη-μέλη έχουν πολύ θετική άποψη όσον αφορά τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και, την προβολή των έργων και όπως βλέπετε ε, εδώ πέρα σε μερικές περιπτώσεις ε, κάποιοι βαθμοί είναι βέβαια πιο χαμηλοί από άλλους φυσιολογικό. Όμω τώρα για να δούμε τι γίνεται με τι σχέσει τράπεζα και κοινοβουλίου. Ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αλλά και η Επιτροπή Οικονομικών Εμπνευστικών Υποθέσεων είναι οι αρμόδιες για τι δραστηριότητε τη Τράπεζα. Και έχουμε αιτήσεις εκθέσει, οπότε έχουμε υψηλό επίπεδο εποπτεία τη ε, ε, ε, και αυτά αποτελούν την αφετηρία για περαιτέρω έλεγχο, αλλά τέλος πάντων η σχέση με την πολιτική συνοχή είναι κάτι το οποίο γίνεται κατά περίπτωση και ad hoc, οπότε βλέπουμε εδώ ότι ο βασικός συνομιλητής της ε, Περιφερειακής Επιτροπής για αυτές τις δραστηριότητες είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί υπάρχει περιορισμένος άμεσος έλεγχος της τράπεζας από ε, την Επιτροπή Περιφερειών. Αυτό όμως δεν οφείλεται σε κάποιο είδους ε, δυστροπία της, ε, της, της τράπεζας. Και βλέπουμε επομένως τι γίνεται για αυτούς τους του περιορισμένου έλεγχο, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί ο διάλογος, αλλά και η ανταλλαγή γνώσης. Τώρα, η συγκρότηση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του ΕΦΣΙ, οδηγεί ε, στο να έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες ε, της ε, τράπεζας από περισσότερες επιτροπές, πέραν αυτών που αναφέραμε. Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι υψηλού επίπεδου οι σχέσεις τράπεζας και επιτροπής, τα αναφέρθηκε και το καταστατικό της τράπεζας, οπότε ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ε, τράπεζας. Επίσης είναι ο βασικός μέτοχος και όσον αφορά το Ταμείο, στο άρθρο 19 του καταστατικού λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται, να οχλείται για οποιοδήποτε θέμα προκύψει για τι δραστηριότητε και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό συντονισμού. Όμω, σύμφωνα με κάποιε συνεντεύξει, λέμε ότι τα, τα προϊόντα δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου ε, τέλο πάντων ένστασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα αλλά να μην του δίνεται ιδέουσα προσοχή. Χωρί να υπάρχει πρόβλημα με τον δανεισμό καθ' αυτό επίση. Ε, οι σχέσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ε, εξελιχθεί σε σημαντικό αριθμό. Θεωρείται και από τι δύο πλευρέ ε, πολύ πολύ θετική αυτή η εξέλιξη και αρχά τη προγραμματική περίοδου 2007-2013 είπαμε ότι έχουμε κάποια χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία έχει ασχοληθεί η Επιτροπή Ρέτζιο και είπαμε ότι η τράπεζα έχει εμπειρία όσον αφορά ε, την εφαρμογή, υλοποίηση αυτών των χρηματοδοτικών, χρηματοοικονομικών εργαλείων. Από την άλλη μεριά υπάρχει καλύτερη κατανόηση του πλευρά τράπεζα για τι πολυπλοκότητε τη ε, πολιτική συνοχή και του πλαισίου αυτή. Στο, στην περίοδο αυτή, 2007-2013, μπορέσαμε να έχουμε ανταλλαγή γνώσεις, ε, περισσότερη κατανόηση και επίσης του, των δυνατοτήτων των διεθνικών οργάνων. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, υπήρχε αυτού του είδους ε, το χάσμα κουλτούρας, πνεύματος που διέπει αυτά τα θεσμικά όργανα, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για περισσότερο ενταλλαγή πληροφοριών και γνώσης. Επίσης, πολλές φορές ε, υπάρχουν κάποιε δυσκολίες αλλά θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα κέντρα που φάζει κάθε θεσμικό όργανο, με την Κομισιόν και με την Τράπεζα ε, και επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις διαφορετικές προτεραιότητες του καθεσμικού οργάνου και επίσης τους στόχους αυτών των πολιτικών του καθεσμικού οργάνου. Στην περίοδο 14-20 τώρα και πέραν του 20 είπαμε ότι το Ταμείο αλλά και η Τράπεζα θα πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα χρηματοδοτικά όργανα. Ακόμα η κατάσταση, το τοπίο είναι ακόμα ξεκάθαρο. Κάποια κράτη-μέλη ακόμα έχουν ισχυρή, στενή εταιρική σχέση με την Τράπεζα και επιδιώκουν στην συνέχεια αυτές τις σχέσεις. Ε, κάποιοι θέλουν να βελτιώσουν, διευρύνουν αυτές τις σχέσεις και σε κάποιε περιπτώσει δεν είχε τόσο σημαντικό ρόλο η τράπεζα, θέλουν να αναβαθμιστεί, α πούμε σε Σουηδία, Νέα Φιλανδία, αλλά και επίση σε κάποιες περιφέρειες που ανήκουν στην Γαλλία. Έχουμε το, την πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εδώ υπάρχουν κάποιες συνέργειες μεταξύ προγραμμάτων υποστήριξης της ε, τράπεζας σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο ενωσιακό και εδώ συνδυάζουμε τους ε, πόρους από διάφορα προγράμματα όπως το COSME, το Horizon 2020 για να χρησιμοποιηθούν, για να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της ε, τράπεζας από τον ιδιωτικό τομέα και από τα εθνικά θεσμικά όργανα. Πάντως η τράπεζα παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διάρθρωση των ε, επιχειρήσεων, των, προγραμμάτων υποστήριξης, ε, όπως ορίζει το άρθρο 39 του σχετικού κανονισμού. Και είπαμε ότι τα κράτη-μέλη που συνεργάζονται θα πρέπει να συνάψουν μια συμφωνία χρηματοδότησης. Οπότε η σχετική πρωτοβουλία όμως ακόμα ε, δεν έχει φτάσει εκεί που θέλουμε. Και έχουν πέντε κρατημέλη, Βουλγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία, προσυπέγραψαν αυτή την πρωτοβουλία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναμένεται και η Φινλανδία να αποφασίσει σχετικά. Όμως, επειδή βάσει των πληροφοριών που έχουμε τώρα, είπαμε ότι έχουμε πρικοδότηση για 1,2 δις, δηλαδή 15% του, ε, της οροφής που προβλέπεται για αυτή την πρωτοβουλία που είναι 8,2 δις. Ε, για να δούμε τώρα, είπαμε ότι το Ταμείο των Επενδύσεων ε, προκάλεσε τον ενδιαφέρον πάρα πολλών επιτροπών του Κοινοβουλίου και της δικής σας επιτροπής. Επίσης, το, η, τράπεζα θα έχει εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, του ΕΦΣΗ, οπότε οποιαδήποτε σχέδια ή προγράμματα θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την τράπεζα. Και έχουμε τις διαδικασίες που διέπουν αυτά τα σχέδια προγράμματα και είπαμε ότι υπάρχουν ε, κάποιοι κανόνες που εξασφαλίζουν το ότι το ΕΦΣΙ θα είναι υπόλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αυτά για την ε, περιφερειακή πολιτική. Έχει το τονίσει η Κομισιόν το ότι είναι συμπληρωματικά το εύση με το έργο της ε, Τράπεζα. Οπότε ο στόχος του εύση είναι αποτελεσματικότητα, όχι ε, δίκαιη κατανομή των πόρων. Αλλά αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι το πώς θα υπάρχει επιλογή των καταλήλων έργων προγραμμάτων χωρίς να παροξύνεται η ανισότητα των περιφερειών. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να κάνει αυτό στην διαλογή το ΕΦΣΙ και θα πρέπει να έρονται οι συγκρούσεις κάποιων ε, κανόνων που διέπουν τη δουλειά αυτών των θεσμικών οργάνων μεταξύ τους. Και τώρα πάλι τις σκητάλια στον, στον Ευχαριστώ. Ας προσπαθήσω λίγο να συνοψίσω ε, τη μελέτη και τα βασικά σημεία να σας αναφέρω. Ε, για την παρουσίαση με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο σημείο είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Ο τρόπος με τον οποίο αυξήθηκε ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην πολιτική συνοχής ε, ξεκίνησε στην αρχή από κάποια τοπικά περιφερειακά δάνεια, μετά επεκτείνεται στάθηκε σε ε, διαχείριση, παροχή συμβουλών, αναλύσεων και δημιουργία δυνατοτήτων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ως πτυχές της πολιτικής συνοχής. Μία από τις ερωτήσεις που έγινε από την αρχή ήταν πόσο αποδίδουν όλες αυτές τις δραστηριότητες της τράπεζας πολιτικής πολιτική Εδώ είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε μια κρίση. Υπάρχουν κάποια ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στα κράτη-μέλη και δείχνουν ότι υπάρχει ψηλού επίπεδου ε, προστιθέμενη αξία ε, ε, στα μάτια των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και επίσης, από διάφορες αξιολογήσεις που έχουν γίνει, φάνηκε ότι αξιολογούνται με μονομένες δράσεις, όπως ο Τζέρεμι και η Τζέσικα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν έχουμε δυνατότητα να έχουμε πλήρη εικόνα της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της πολιτικής συνοχής. Αυτό με τη σειρά του δυσχεραίνει την πλήρη εκτίμηση, ακόμα και την πλήρη κατανόηση της κατάστασης. To address um, the accountability transparency. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ε, λογοδοσία, την ε, διαφάνεια και την ε, ορατότητα και την προβολή, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να βελτιώσει όλες αυτές τις πτυχές και αυτό φαίνεται στη μελέτη που έγινε στα κράτη-μέλη και σε πολλαπλό βαθμό. Ωστόσο υπάρχει ακόμα πολλής χώρος για βελτίωση και μεγάλη ανάγκη θα πρότεινα της κατανόησης με πιο συστηματική αξιολόγηση μετά από πιο συστηματικές εκθέσεις και πιο συστηματικό έλεγχο. Χρειάζεται περισσότερη μέθοδος. Γι' αυτό κάνουμε και συστάσεις εμείς στην έκθεσή μας που εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες. Μπορούν να ξενοποιηθούν πρώτον ο έλεγχος και το δεύτερο η καλύτερη κατανόηση της ε, δράσης. Ε, σε ό,τι αφορά τον επίσημο έλεγχο τώρα, ε, τι ζητούμε και τι συστήνουμε μάλλον το Κοινοβούλιο δια της Επιτροπής σας ε, θα μπορούσε να υποστηρίξει και να προωθήσει περισσότερη λογοδοσία για το ρόλο ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βλέπουμε και την ε, γνωμοδότηση του 2015 και ζητάμε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα κεφάλαιο, ένα παράρτημα για την πολιτική συνοχής στην ετήσια έκθεση ε, ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ακριβώς για να βελτιωθεί η εφαρμογή και η υλοποίηση των στόχων της πολιτικής συνοχής. Πέρα από τον επίσημο έλεγχο υπάρχει και πολλής χώρος για την καλύτερη κατανόηση και την πρόθεση το τι ε, κάνει, ποιες είναι οι δραστηριότητες της τράπεζας με περισσότερο διάλογο και μάλιστα μόνιμο και διαρκή μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της τραπέζης της ίδιας για να υπάρχει καλύτερη αμοιβαία κατανόηση της συνεισφοράς του καθενός στην πολιτική συνοχή. Η σχέση με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ενισχυθεί με διάφορα μέτρα και σε πολιτικό επίπεδο και της Επιτροπής ε, να πηγαίνει η Επιτροπή σας στην Τράπεζα Επενδύσεων όπως πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ε, να έχουμε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής έκθεση πεπραγμένων προς την Επιτροπή σας από πλευράς της Τράπεζας. Τρίτον, σεμινάρια και ε, εργαστήρια σε διοικητικό επίπεδο για να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και να υπάρχει μεγαλύτερη προβολή και ορατότητα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και να υπάρχει καλή και αγαστή διοργανική συνεργασία. Ε, πιο λεπτομερείς μελέτες επίσης για συγκεκριμένα στοιχεία εφαρμογής πολιτικής συνοχής και επίσης η ε, πρόσληψη προσωπικού από άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν γνώση για να μπορέσει αυτή να μεταλαμπαδευτεί και στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέλος έκθεση ιδίας πρωτοβουλία που θα συμπεριλαμβάνει και το ρόλο της τραπέζης ε, στην πολιτική σύνοχη. Τέλος, παραδοσιακά οι πανεπιστημιακοί ζητούν περισσότερη έρευνα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, υπάρχουν πραγματικά τομείς σημαντικοί που χρειάζεται περισσότερη έρευνα και περισσότερη συζήτηση για να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα και κενά που έχουμε ως προς τη γνώση μας. Άρα χρειάζεται περισσότερη έρευνα και ιδιαίτερα επιτροπή σα, αλλά και γενικότερα το Κοινοβούλιο και ο πανεπιστημιακό κόσμος και η πανεπιστημιακή κοινότητα, μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει τη δέουσα προσοχή και δεν έχουν δώσει την ίδια προσοχή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, όσο σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ε, ειδικά λοιπόν εμεί ε, ζητούμε να διερευνηθεί περισσότερο ο ρόλος τη ΕΤΕ στην εφαρμογή των προγραμμάτων τη πολιτική συνοχή στα διάφορα στάδια, το στάδιο του προγραμματισμού, της δρομολόγησης, της δημιουργίας έργων, ε, λεξιμότητα, διαδικασία επιλογής ε, των ε, έργων, να γίνει περισσότερη έρευνα για τις δανειοδοτικές δραστηριότητες, χορηγήσεις που κάνει η τράπεζα, ιδιαίτερα οι δραστηριότητε lending και blending στην πολιτική συνοχή και πώς συνεισφέρουν σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής. Και ένα τελευταίο που προτείνουμε ως μελλοντική έρευνα, επειδή αλλάζει το σκηνικό τώρα και τα δεδομένα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, πρέπει να δούμε τη νέα κατάσταση και θα υπάρξει μια μόνιμη ανάγκη, όχι μόνο να το παρακολουθούμε αυτό, αλλά και να ερευνούμε το ρόλο και τον αντίκτυπο που θα έχει το ΕΦΣΙ στην πολιτική συνοχή σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank you. Εμείς σας ευχαριστούμε για την τόσο λεπτομερή παρουσίαση και ενημέρωση που μας κάνατε. Ε, ανοίγει τώρα η συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Έχω ήδη ένα όνομα. Ε, την κυρία Μάλετιτς και μετά ο κύριος Βανίστερ ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι οι συστάσεις σας είναι έξοχες. Σας ευχαριστώ για τη μελέτη. Μ' αρέσει που βλέπω ότι διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάλυση της κατάστασης επικρατή στα κράτη-μέλη, να αυξηθεί η ορατότητα των δραστηριοτήτων της ΕΤΕ και χρειάστηκε συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στις δραστηριότητες της ΕΤΕ. είπατε ότι δεν υπάρχει έλεγχος και επισκόπηση της τη πολιτικής συνοχής και των σχετικών έργων. Αυτό με εξέπληξε, αυτό χρειαζόμαστε. Και χρειαζόμαστε και κάτι παραπάνω. Όταν μιλάμε για πολιτική συνοχής, αναφερόμαστε στην ανάγκη καλύτερου συσχετισμού και συντονισμού της πολιτικής συνοχής με την περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική μεταφορών, ενεργειακή πολιτική, ανάπτυξη πέθρου, αστική πολιτική, έρευνα, καινοτομία, αναπτυξιακή πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΤΕΘ στην υλοποίηση όλων των πολιτικών. Αυτό πρέπει να αναλυθεί. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη κάθε κράτους μέλους Δύο uh, στα πλαίσια οικονομικής πολιτικής και περιορισμού των ελλημάτων των κρατών μελών, διότι δανειοδοτείεται και τα δάνεια ε, απορροφούνται στο δημόσιο έλλειμμα. Και καμιά φορά τα χρήματα πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται συντονισμό σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Θα πιάσουν τόπο τα χρήματα που δίνεται στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται συντονισμός και συσχετισμός με τις οικονομικές πολιτικές. Σημαντικότατο στοιχείο. Αναφερόμενοι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πήραν εγγυήσεις από την ΕΤΕ αλλά δεν μπορούσαν τελικά να πάρουν το δάνειο λόγω των οικονομικών συνθήκων στη χώρα, λόγω κατεκαιρματισμού της αγοράς. Και ο ρόλος της ΕΤΕ είναι να περιορίζει τον κατεκαιρματισμό της αγοράς. Και να είναι ισότιμες συνθήκες δανειοδότης στα διάφορα κράτη-μέλη. πήραν την, είχαν την εγγύηση πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν το δάνειο στην πράξη λόγω τη καταστάσεως συγκεκριμένου κράτου μέλους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να δούμε. Να μπορεί να εμπλέκεται στι διάφορε αγορέ πιο άμεσα η ΕΤΕ. Ευχαριστώ ο Βαν Νίστελ Ρόι. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, ε, τόσο βαριά ημερήσια διάταξη και τόσο σημαντικό θέμα στο μενού μας, να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και πώς να τα συνδυάσουμε αυτά με την κανονική μας δουλειά. Γιατί μας έπεσαν βαριά όλα αυτά που ακούσαμε. Είναι πάρα πολλά για να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε και να τα χωνέψουμε και να τα βάλουμε στη δουλειά μας. Ακούγοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη λένε κάθε μέρα ε, και το Twitter του κύριου Κατάινεν Όλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ, το ΕΦΣΙ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε μέρα τα ίδια να μασούν και μερικάζουν και είναι της μόδα τώρα αυτό τον καιρό ε, οι αναφορές. Ε, όταν δίνουν επιδοτήσεις σε έργα, λέει αυτό τελείωσε, τώρα πάμε στα δάνεια. Δεν ξέρω, μήπως είναι στρεβλή αντίληψη που έχω. Όταν ακούω όμως αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό αντιλαμβάνομαι. Και μπορεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει αργότερα, ξέρω εγώ, την ε, έκθεση και αυτά που ακούσαμε τη μελέτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι θα συζητούμε σήμερα αυτά τα θέματα. Τώρα, μια που μιλάμε για τη σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι μυστήρια η σχέση μας γιατί είναι λίγο κράτος εν κράτη. Άκουσα προσεκτικά ε, τις συζητήσεις που έγιναν και για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ήταν ότι εμείς είμαστε αρμόδιοι. Εγώ έχω κάνει γνωμοδότηση για το ΕΦΣΥ και είπαμε θα πρέπει να βρούμε πώς λειτουργεί ο καθένας και ποια είναι η θέση του καθενός. Και μας είπαν ότι είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και περίπου μην ανακατεύεστε εσείς, έτσι. Εκείνοι έχουν την αρμοδιότητα, έχουν το Διοικητικό Συμβούλιο, τους εμπειρογνώμονες, κάτω τα πολιτικά σας χέρια από αυτό το πράγμα. Και τώρα έρχεστε και μας λέτε ότι να τα φτιάξουμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα Επενδύσεων ότι δεν είναι τόσο σαφής η σχέση. Μα θέ μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι από έτσι, από την αρχιτεκτονική. Συζητούμε στο άρθρο 63 φέτος την αντίστοιχη έκθεση για τις επιδόσεις. Δεν συζητούμε όμως με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα που μας φέρατε εδώ για τη λογοδοσία για τη διαφάνεια, για την προβολή, για την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πού είναι αυτή η σχέση. Μήπως είναι λίγο διαφορετική και λίγο πιο μυστήρια. Και αν θέλουμε να έχουμε τον ίδιο έλεγχο, θα είχα και εγώ να προσθέσω διάφορα πράγματα. Συνεργάζομαι με την αντιπροσωπεία, μάλλον πήγαμε στη Σεβίλη, στην Ανταλουσία, στην περιφέρεια εκεί, με τη Ρέγγι. 400 εκατομμύρια ευρώ έχουν χαθεί σε ένα από αυτά τα προγράμματα με τον Τζέι, Τζέρεμι, Τζέσικα, δεν ξέρω, εξαφανίστηκαν. Έκαναν φτερά. Τόσο καλύτερη πια είναι η διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από ό,τι φαίνεται όχι. Οπότε κάτι πάει στραβά εκεί, έτσι. Και θα πρέπει να τα συζητούμε και αυτά με την ΕΤΕ. Δεν τα συζητούμε στην ημερήσια διάταξή μας, δεν είναι τακτική επαφή και έχετε δίκιο. Ότι θα πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα. Κάπως έχουμε αποστασιοποιηθεί, έχουμε απομακρυνθεί από το δικό μας ρόλο που είναι ε, ο έλεγχος της συνοχής και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και ξέρω ότι υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που βάζει χοντρά λεφτά ε, στα Ταμείο Συνοχής για αυτοκινητοδρόμους, ιδιαίτερα στις χώρες συνοχής. Εδώ δεν βλέπω τίποτα να λέτε γι' αυτό. Εκεί να δείτε κονδύλια και πόσο σημαντικά είναι και πόσο ενέχονται σε αυτές τις πολιτικές. Αυτό που χάθηκε. Και κάτι που είπατε για την αργή απορρόφηση και ε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν κάποιος πρέπει να το ξέρει εσείς θα είστε αυτοί αφού το μελετήσατε. Αυτό γιατί συμβαίνει. είναι αργή σε σχέση με προηγούμενους καιρούς, προηγούμενες περιόδους ή γιατί έχει αλλάξει αγορά και δεν τα απορροφά. Ξέρετε ότι τα επιτόκια έχουν πέσει κατακόρυφα για τα δάνεια. Αν αρχίζει να διαπραγματεύεσαι με την ΕΤΕ το πρώτο έτος ή το δεύτερο έτος, είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Θα πάρεις δάνειο, γιατί στην αγορά έχει πέσει, ε, έχουν πέσει τα επιτόκια. Αυτά ακούω. ότι είναι πολύ ψηλά τα επιτόκια και δεν είναι αγωνιστικά της αγοράς. αυτό ακούμε ως σχόλια. Για πού είναι τα θετικά για την πολιτική συνοχή και η χειρονομία που θέλει να κάνει η Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν καταλαβαίνω αυτό γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σας και γιατί δεν απορροφώνται τα δάνεια. Θα μπορούσατε λίγο να μας διαφωτίσετε περισσότερο. Γενικά έχω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ήρθε αυτή η μελέτη και η εκθεσή και να της ε, συντονίσουμε ε, με άλλες ε, συζητήσεις που έχουμε προγραμματίσει στην Επιτροπή μας για τη νέα περίοδο, ας πούμε, η έκθεση για το άρθρο 60 εδάφιο 3 και να δούμε και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ κρατών. Πολύ συχνά δεν έχει υποχρέωση κάποιος να το κάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ας πούμε, είναι στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν. Δεν είναι κουστούμι που ράβουμε για όλους. Μπορεί να είναι κάθε φορά στα μέτρα της μιας χώρας ή της άλλης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ πάντως για αυτή τη μελέτη. Και είναι και θεμελιώδη αυτά τα πράγματα και πάρα πολύ βασικά. Και αν ακολουθήσουμε τη γραμμή αυτή που λέτε ότι η δική μας Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα ηγηθεί, ελπίζω να ακολουθήσουν την υπόδειξή σας αυτή ε, και οι άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Εγώ μαζί σας είμαι μέχρι τέλους, διότι θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο ε, σημαντικό αυτό, αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα τα επόμενα χρόνια, αν καταλάβει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιδείξει ότι τρέχει και τα διαχειριστεί σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταμάτο ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Και μετά η κυρία Βάνα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Όλοι οι συνάδελφοί μας θέλουμε να μελετήσουμε λεπτομερέστερα την έκθεση. Το Κοινοβούλιο αντιμετώπισε σημαντικό κόστος 43 εκατομμύρια ευρώ για να... χιλιάδες ευρώ μάλλον για να αναπτυχθεί. Ακούγοντας λοιπόν την παρουσίασή σας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει, υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος των παρεμβάσεων. Ξεκινώντας και από τον ορισμό των κριτηρίων για τον καθορισμό των έργων, ούτως ώστε να αξιολογείται και ποια είναι η επιρροή όσον αφορά την πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βλέπουμε στον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των διαφόρων χρηματοδοτήσεων για τα έργα. Θα σταθώ σε διάφορα προγράμματα που παρουσιάζουν κάποια κράτη-μέλη προς από την ΕΤΕ και από το ΕΦΣΙ. Έχω την εντύπωση ότι πολλές από τις αιτήσει στρέφονται προς το παρελθόν με την υποστήριξη στις ορυχτές πηγές αέριο, φυσικό αέριο, αποθήκευση και αυτή και τη δίληση του πετρελαίου, ε, το ε, έλαιο, δηληστήρια παλαιάς τεχνολογίας. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μου κυρίως. Λοιπόν, η αγωγοί χρειάζονται επιλογές και μπορεί να επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον. επιλογές που γίνονται καυστήρες και αντιδραστήρες και λοιπά είναι επιβλαβείς ε, για το περιβάλλον και θα πρέπει επενδύσεις να έχουν στόχο την κυκλική οικονομία. Ερώτηση. Για τον προγραμματισμό αυτό η ΕΤΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα συνεχίσουν συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των διαφόρων μέσων που θα είναι εναλλακτικά και θα συμπληρώνουν τις παραδοσιακές χρηματοδοτήσεις. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα, θα είναι δημιουργη... Θα, μήπως θα αυξάνεται το κίνδυνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Να ήθελα να επενθυμίσω και στους συναδέλφους ότι το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο συνέστην την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα τακτικό έλεγχο και τη χρήση δικτών επιδόσεων που θα μπορούν να συγκρίσιμοι μεταξύ κρατών μελών και αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να ισχύσει και για την ΕΤΕ. Εν κατακλείδη, θα ήταν καλό κατά την άποψή μα και κατά την άποψή σα, μάλλον να ξεκινήσουμε έναν έλεγχο με μια αξιολόγηση ομοιογενή, με μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την επιλογή των έργων που θα είναι μακροπνού εμπνεύσεως για τη συνοχή και υπέρ της υγείας του περιβάλλοντος και υπέρ της ζωής θετικά, θετικές επιλογές για τη ζωή όλων των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ η κυρία Βάνα που θα είναι η τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Αυτό που θέλω να πω είναι σχετικό με αυτό που είπε η κυρία Λέω Όταν πιάνουν τόπο τα χρήματα αυτά τα πιθανέ τράπεζα και τι γίνεται με τα ουσιαστικά αποτελέσματα. Μήπω θα μπορούσατε να μα πείτε δύο λόγια παραπάνω, να μα εξηγήσετε ακριβώ πώ η τράπεζα ε, συνεισφέρει στην επιτεύξη των στόχων του Horizon 2020. Ας πούμε, πέστε μας ε, τι γίνεται όσον αφορά την οικονομική κοινωνική συνοχή, κάποια δηλαδή αριθμητικά στοιχεία ε, μήπως έχετε και κάποια στοιχεία για την παιδεία, για την αλλαγή του κλίματος, ε, για την αγορά εργασίας, γιατί είναι, είναι το θέμα του τι, τι, τι νούμερα ε, ε έχει αυτή η ιστορία και όχι μόνο το τι ποιότητα ε, προκύπτει από, τα, από, την συμβολή της τράπεζας. Δηλαδή θέλω να δούμε ακριβώς ποια είναι τα, τα, συνολικά ποσά που προκύπτουν. Και έτσι μπορούμε να αξιολογήσουμε και τι γίνεται σε σχέση με τους στόχους ενώπιση του 2020 και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον να δώσουμε ε, τον λόγο στον ε, κύριο Τόμας Δεμπέτον που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν πρόφερα σωστά το όνομά σας. Ε, περίπου. Μήπως θέλετε το λόγο. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. πολλές οι ερωτήσεις και φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε λάβει αυτό το, το σχέδιο της μελέτη πριν από τρεις μέρες οπότε και, και εμείς δεν είχαμε το χρόνο να δούμε τις λεπτομέρειες και πριν από τρεις εβδομάδες επομένως είχαμε ε, την ευκαιρία να δούμε αυτά τα κεφάλαια αλλά δεν μπορέσαμε να δούμε συμπεράσματα και συστάσεις πιο νωρίς οπότε δύσκολο τώρα να σας πω τα σχετικά πάντως από την εισήγηση που άκουσα μπορούμε να σας πούμε ότι αναγνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε να επιλύσουμε σε σχέση με την συνεργασία, ε, σε σχέση με ε, τις εργασίες της Τράπεζας Εργασίας. Πάντως ε, για τα θετικά που ακούσαμε, Τζέσικα, Τζέρεμι, για την καινούργια πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ, όλα αυτά αφορούν την υπόθεση της διαχείρισης, ούτως ώστε να αναπτύξουμε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάποιου είδου ε, άλλα έργα, προγράμματα που έχουν σχέση με τα Ταμεία Συνοχής και επίσης με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οπότε, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να ξαναμελετήσουμε τα στοιχεία και θα σας ε, σχολιάσουμε τις ε, συστάσεις εν ευθέτω χρόνο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ελπίζω ότι όταν τα ξαναπούμε θα έχετε να μας πείτε περισσότερα. Γιατί εδώ στην Επιτροπή μας θα κάνουμε μια συνεδρίαση όπου θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα πλαίσια του ελεγκτικού μας ρόλου. Οπότε οι εκπρόσωποι της τράπεζας θα είναι εδώ ε, επίσης θα είναι εδώ οι διαχειριστές του Εύση και επομένως ε, τότε περιμένουμε να μας πείτε περισσότερα. Κύριε Μπάχτερ, καθηγητά, θέλετε να απαντήσετε τις υποβληθείς ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Μάλιστα ευχαριστώ πολύ για τα όσα ερωτήσατε και για τα όσα σχολιάσατε. Οπότε για να δούμε και ως απόφατα συμπληρώσει ο συνάδελφος. Πρώτη ερώτηση. Όσον αφορά αυτό το οποίο σας ανέφερα για τον ρόλο της τράπεζας για διάφορες πολιτικές και για το Horizon 2020. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, γιατί εδώ έμεσα υπάρχει επίδραση στην πολιτική συνοχής. Έχουμε επίσης το Connecting Europe Facility, το COSME, το πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης γνωρίζουμε ότι έχει σημαντικό ρόλο η τράπεζα. Όμως δεν έχουμε συλλάβει το μέγεθος της ε, επίπτωσης του ρόλου της ε, τράπεζας και αυτό είναι το απογοητευτικό στοιχείο. Ξέρουμε κάποια στοιχεία, αλλά δεν έχουμε ακόμη ε, εικόνα του συνόλου του τοπίου, των επιπτώσεων του έργου της τράπεζας. Οπότε, με τις εγγύσεις, με τα δάνεια και όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται που είναι σημαντικό γιατί σχετίζει με αυτό που και ο Φαν Νίστελ Μα είπε και αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία σε σχέση με τα δάνεια και τις ενισχύσεις, grants. Θα πρέπει να γίνει ένας απολογισμός, μια καταγραφή τέλο πάντων του τι έχουμε κάνει και πού έχουμε φτάσει όσον αφορά τα αποτελέσματα την αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων χρηματοδότησης. Άρα, δεν πρόκειται για πανάκια. αυτή η χρηματοδότηση είχε επικουρικό χαρακτήρα, δεν υποκαθιστά τις ενισχύσεις. Άρα, αυτού, αυτά τα δάνεια της τράπεζας πρέπει να τα χρησιμοποιούμε παράλληλα με τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και ενισχύσεις. Σε σχέση με δυνατότητες διοικητικές και σε σχέση με κάποιους δικαιούχους. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για την αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων είναι το πώς θα γίνει η υλοποίηση μέσα σε ένα περιβάλλον συμβούλων κλπ. Άρα επομένως έχει σημασία η συγκυρία το περιβάλλον, αν θέλετε, της ε, εφαρμογής, της υλοποίησης. Η ποιότητα των επιλεγέντων σχεδίων προγραμμάτων έχει σχέση με την αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουμε. Οπότε και προκύπτει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ε, εφαρμογή αυτών των χρηματοοικονομικών εργαλείων που χρησιμοποιεί η τράπεζα. Έχουμε από τη μία μεριά τους εμπορικούς στόχους της τράπεζας. Και από την άλλη μεριά έχουμε τους στόχους που τάσει η περιφερειακή πολιτική ή πολιτική συνοχής. Οπότε θα πρέπει οι επιμέρους ε, αντιφάσεις, ε, συγκρούσεις θα πρέπει να αρθούν. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο σε συγκυρία οικονομικής κρίσης. Άρα δεν είναι σαφές κατά πόσον οι στόχοι πάντοτε κυριαρχούν σε αυτές τις συγκρούσεις. Απ' την άλλη μεριά όσον αφορά τον διαρχή έλεγχο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες, κάποια στοιχεία δεδομένα για το πώς τα χρηματοδοτικά όργανα θα βοηθάνε σε παραγωγικότητα, απασχόληση και ανοτομία. Δεν ξέρουμε εάν ε, τηρούνται οι προσδοκίες που υπάρχουν από αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί όλα αυτά είναι σχετικά πρόσφατα ε, όργανα, πρόσφατα εργαλεία μάλλον, τα οποία μας προέγυψαν. Ο συνάδελφος να μπορεί να συνεχίσει. Ευχαριστώ, Τζον. Να προσθέσω το εξής για την ερώτηση του κύριου Φαν όσον αφορά για τις ΜΜΕ, όσον αφορά το χαμηλότερο από τις προσδοκίες επίπεδο απορρόφησης. Γιατί έχουμε εδώ πολλές πιθανές εξήγησεις. Οπότε εδώ πέρα προκύπτει ότι ίσως χάνεται ο έλεγχος όσον αφορά το πού πάει αυτή η χρηματοδότηση τι απογίνεται αυτή η χρηματοδότηση. Ίσως αυτό εξηγεί, ίσως και εν μέρει, το γιατί έχουμε χαμηλότερη απορρόφηση. Επίσης, έχουμε το άρθρο 59 του κανονισμού. Αυτό θεσπίστηκε σχετικά αργά, κατόπιν και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Οπότε η κατανομή των πόρων σε εθνικό επίπεδο ήδη είχε προχωρήσει. Ήδη είχαν ληφθεί οι σχετικέ αποφάσεις, οπότε απαιτεί αυτή η πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα και κατόπιν αναπρογραμματισμό της κατανομής των πόρων, οπότε προκύπτουν πολλά προβλήματα πολιτικά σε πολλές περιπτώσεις, άρα έτσι να δείτε το τι απογίνονται αυτά τα 1,2 δις Βέβαια άλλαξε η οικονομική συγκυρία σε κάποιες χώρες. Δεν γίναν τα πράγματα έτσι όπως τα περιμέναμε στην αρχή. Άρα υπάρχουν πολλές εξηγήσεις γι' αυτό που είπατε. Αλλά ακριβώς η συγκυρία κατά πολύ καθορίζει ότι γίνεται. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε για την σημερινή σας παρουσίαση. Ευχαριστώ για αυτή την μελέτη. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να αναλύσουμε αυτή την έκθεση και ελπίζω να διεξαχθούν καρποφόρες συνομιλίες με την ΕΤΕ στην επόμενη επίσκεψή της στην Επιτροπή μας. Θα γίνει στο μέλλον αυτή η συνάντηση. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης μακροπεριφερειακή στρατηγική στην περιοχή των Άλπαιων στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπως για τη Βαλτική, τον Δούναβη και την περιοχή της Αδριατικής είναι σημαντικό στοιχείο για το σχεδιασμό της εδαφικής ε, συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 28 Ιουλίου πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε σχετική ανακοίνωση κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013 ούτως ώστε να συντάξει μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την περιοχή των Άλπαιων. Η στρατηγική θα καλύψει τρεις θεματικές πολιτικές, οικονομική ανάπτυξη, κινητικότητα και συνδεσιμότητα, περιβάλλον και ενέργεια. Στις 17 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή μας αποφάσισε να συντάξει μία έκθεση πρωτοβουλίας νομοθετικού περιεχομένου για, την, ε, το θέμα αυτό. Η κυρία Μπρεσό, η συγγήτρια, θα μας παρουσιάσει τις σκέψεις της, θα παρουσιάσει το σχέδιο εκθέσεως τον μήνα Απρίλιο και πιθανότατα θα ψηφίσουμε τον Ιούνιο την έκθεση στην τελική της μορφή. Έχουμε μέχρι τις 5 η ώρα περίπου στη διάθεσή μας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπρεσό για να παρουσιάσει τις αρχικές της απόψεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως υπενθυμίσατε, η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε το 2011 για την περιοχή των Άλπαιων και στο Δεκέμβριο του 2013 ανεκρίθη η Επιτροπή του 2015 παρουσίασε σχέδιο δράσεως και πρόσφατα το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε πλέον αυτή την πολιτική και δρομολογήθηκε επίσημα στη Σλοβενία τις 25 και 26 Ιανουαρίου και όπως υπενθυμίστηκε είναι η τέταρτη μακροπεριφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι όλοι μας θυμόμαστε τον Δούναβη, τη Βαλτική, Αδριατική Ιωνίου, τις άλλες πρωτοβουλίες. Η στρατηγική μακροπεριφερειακή δημιουργήθηκε κυρίως από πρωτοβουλίες διακυβερνητικής φύσεως. Σε περιοχές της Υπήρου μας που είχαν διαιρεθεί, είχαν διχαστεί από σιδηρά παραπετάσματα και πολέμους και θέλαμε να υπάρξει συνεργασία θεσμική και οικονομική μεταξύ των διαφόρων αυτών περιοχών κατέστησαν δυνατές μέσω της συνθήκης της Λισαβόνα. με στόχο την εδαφική συνοχή. Πιστεύω ότι είναι μια καλή έκφραση αυτής, του στόχου της εδαφικής συνοχής αυτές οι πρωτοβουλίες και θα πρέπει να καθοριστεί αυτή η πολιτική εδαφική συνοχής και να γίνει πιο καλά κατανοητή ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Νομίζω ότι σήμερα για την ανάπτυξη των πρωτοβουλίων αυτών και για περαιτέρω τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει να ενταχθούν καλύτερα στην κοινοτική μέθοδο διότι ε, δημιουργούνται μέσω διακυβερνητικής μεθόδου και εγκρίνονται σε επίπεδο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Χρειάζεται διαφορετική μέθοδος. Είναι διαφορετική μέθοδος από την κανονική μέθοδο θέσπισης νομοθεσίας. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό που υπάρχει εκεί όσον αφορά το στρατηγικό προγραμματισμό κάτωθεν εν συγκρίση με όλες τις προσπάθειες που κατευλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει, ήταν μέσα άνωθεν επιβαλλόμενα. Καθοριζόταν εδαφικές στρατηγικές άνωθεν όμως προερχόμενες. Εδώ για πρώτη φορά το όλο εγχείρημα κάτωθεν κινείται. Και είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτή την προσέγγιση, να αξιοποιήσουμε αυτό που θα ήταν αναγκαίο για να αντιμετωπιστούν και θεσμικά προβλήματα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από την αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την αρχή της δρομολογήσεως μακροπεριφερειακής στρατηγικής και στην φάση του προγραμματισμού που το κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό γίνεται ήδη, αλλά και μετά στην εφαρμογή, υλοποίηση και συντονισμό με άλλες στρατηγικές πρέπει να συμμετέχει περισσότερο και γενικότερα. Αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να εντάσσονται στην πολιτική εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα χρειαζόταν επίσης και επίσημη εμπλοκή του Ευρωκοινοβουλίου στο μέλλον με το ρόλο συνομοθέτου που διθέτει και στην αρχική δρομολόγηση και στην έγκριση και στον έλεγχο των αποτελεσμάτων που επιτυχάνονται. Στατηγικές για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι πάρα πολύ σημαντικές που αφορά περίπου, είναι περίπου 300 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι θέσεις στρατηγικές καλύπτουν περίπου 300 εκατομμύρια πολίτες. Άρα, αφορούν μελλοντικό χρήσο και των διαφόρων πόρων της Ένωσης. Τεράστια ανάπτυξη. Θα πρέπει να ελέγχεται πιο άμεσα από τους εκλεγμένους ε, εκπροσώπους του λαού. Όπως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί δημοκρατικά τους πολίτες. Χρειάζεται προβληματισμός από αυτού. Διαφορετικός καθορισμός των διαδικασιών, καλύτερος συντονισμός με άλλες πολιτικές της Ένωσης. Και διότι θα υπάρξουν και άλλες προτάσεις, χρειάζεται νομοθετική πράξη που θα καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου, που θα κινούμαστε και στο μέλλον, αλλά και που θα ε, κινούνται και ήδη δρομολογηθήσεις ε, προσπάθειες. Θέλουμε λοιπόν καλύτερη πλησίωση των κάτω ε, κινουμένων τέτοιων πρωτοβουλίων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την επικουρικότητα. Μέχρι τώρα, ο ρόλος της προώθησης ε, ανήκε στις εθνικές αρχές και στις κινητικές αρχές που εκαλούνται να συμμετάσχουν από τι εθνικέ αρχέ, όμω πιστεύω ότι αυτό ο ρόλο πρέπει να είναι πιο συγκροτημένο από την αρχή και η πραγματική διακυβέρνηση των προγραμμάτων, συνοποίηση των προγραμμάτων, θα πρέπει να αφορά τοπική αυτοδίκηση, που πρέπει να πρωταγωνιστεί στην εδαφική αναπτυξιακή πολιτική. Διαφορετικά, οι πρωτεύουσε των κρατών είναι πάντα μακριά από την τοπική αυτοδίκηση. Και τέτοιες σημαντικές προσπάθειες να μην υλοποιούνται σωστά, με συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα είναι κρίμα. Και σε κάποια φάση πρέπει να το αναλύσουμε και εμείς στην Επιτροπή μας. Και όταν κάνουμε τις αξιολογήσεις των διαφόρων στατικικών. Η στατικική των Άλπαιων τώρα λαμβάνει η χώρα σε ένα περίπλοκο πλαίσιο. Ε, πολλαπλές συνεργασίες υπάρχουν στην περιοχή. Η περιοχή των Άλπαιων, η Σύμβαση των Άλπαιων, διάφορα προγράμματα Interreg, διάφορες, ε, διάφορες ομάδες συνεργασίας. Είναι ιστορικός χώρος συνεργασίας αυτός. Εκεί είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τη δική μας στατικική και τις ορεινές περιοχές των Άλπαιων, και τις ζώνες γύρω στις Άλπεις αλλά και μεγάλες πόλεις. Αυτές οι περιοχές αντιπροσωπεύουν και οι πόλεις και οι περιφέρειες τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές, από τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που αφορά 70-80 εκατομμύρια άτομα. Υπάρχουν διαφορετικές αξιολογίες στον τον πληθυσμό που καλύπτεται. Άρα αντιμετωπίζουμε μεγάλη περιοχή που μπορεί να επανεξορροπήσει τις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Και έχουμε και σημαντικές οικονομικές περιοχές στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν πρέπει να λησμονούμε και τις ορεινές περιοχές. Ορεινές περιοχές αλλά εμπλέκονται και σημαντικές αστικές περιοχές στο όλο πλαίσιο. Πρέπει να λάβουμε τις δύο πτυχές, δύο όψεις στρατηγικής. Ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ περίπλοκα προβλήματα, αλλαγή του κλίματος Φερρυπίν, που επηρεάζει πάρα πολύ. Και μετά τις παιδιάδες. Εκεί έχουμε δυνατότητες και ανάπτυξης, αλλά και προβλήματα. Είναι περιοχές κυρίως παραγωγικές και βιομηχανικές και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι βιομηχανικές περιοχές στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι σήμερα δεν μπορούμε να αναλύσουμε λεπτομερώς τους τρεις πυλώνες που προτείνονται. Στόχος εκθέσεώς μου θα είναι ο εξής. Να δούμε ποια είναι η θεσμική αρχιτεκτονική. Να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα που δίδεται στις περιφέρειες και στις, στους εδαφικούς φορείς που ήθελαν μια τέτοια στρατηγική. Μετά από τους τρεις πυλώνες που είναι η βελτίωση ανταγωνιστικότητας της ευημερία και της συνοχής της περιοχής των Άλπαιων προσβασιμότητα, διασύνδεσιμότητα που είναι τεράστια προβλήματα διότι η συνδεσιμότητα είναι πολύ δύσκολη. Και δημιουργούνται προβλήματα επαφών και τηλεπικοινωνιών, διασυνδέσεις του διαδικτύου κλπ, ενεργειακές διασυνδέσεις είναι προβληματικές. Και αν λυθούν αυτά τα προβλήματα έχουμε βελτιώσεις οικονομικές. Πολύ σημαντικές στοιχείες λοιπόν. Τρίτο, πτυχίο. Πρέπει να προστατεύσουμε και τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους. Το οικοσύστημα των Άλπαιων, που είναι υπέροχο, από πάντα υπήρχε πληθυσμός εκεί. Από τους πρώτους πληθυσμούς είχαμε εκεί της Ευρώπης που ζούσαν εκεί στις ορεινές περιοχές, στις περιοχές των Άλπαιων και γύρω από τις Άλπεις. Και αυτός είναι πυλώνα σημαντικότατος. Τρεις πυλώνες λοιπόν ανέφερα δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό από την αρχή. Τι θέλουν οι περιοχές αυτές. Να αξιολογήσουμε το εξής. Για να υπάρξει ανάπτυξη και εξελίξεις που ζητήθηκαν. Πώς θα διαμορφώσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές στο σύνολό τους. Δεν χρειάζεται να διατεθούν περισσότεροι πόροι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα για την περιφερειακή πολιτική και άλλες πολιτικές και άλλα προγράμματα που ήδη υπάρχουν όπως για την έρευνα, την ενέργεια, για τη γεωργία τόσες δραστηριότητε ότι αυτές, όλα αυτά να έχουν καλύτερη στόχευση και να καλύπτουν τις ανάγκες περιοχών με ιδιαιτερότητες που δεν εξαρτώνται μόνο από οικονομικές εξελίξεις, καθυστέρηση κλπ. Και δεν έχουν προβλήματα που αφορούν μόνο την οικονομική συνοχή, αλλά έχουν διαθετικά προβλήματα που δεν μπορούν να αλλάξουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά μπορούν να ληφθούν υπόψη στις παρεμβάσεις. Και αν δεν υπάρχουν πρόσθετοι πόροι που διατίθενται, παρόλα αυτά όμως, μπορούν, μπορεί να γίνεται καλύτερη στόχευση μέσω καλύτερης χρήσης των υφισταμένων πόρων που θα καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες. Με βλέπετε με στραβό μάτι βλέπω, ήθελα τα αναφέρω αυτά ξέρετε. Μου λέτε μάλλον ότι πρέπει να σταματήσω. Άρα δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες. Πιστεύω όμως ότι είναι μια ευκαιρία αυτή. Ευκαιρία για προβληματισμό να δούμε πώς οι μακροπεριφερειακές στατηγικές θα εδράζονται καλύτερα στις περιφερειακές πολιτικές και τις πιο γενικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να μην είναι μεγάλα όμορφα λουλούδια που ανθούν και που μαραίνονται πολύ γρήγορα διότι δεν τα ποτίζουμε τα φυτά αυτά, χρειάζεται συνεχής προσοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών, των εδαφικών πολιτικών και να συμμορφώνται με τα αποφασιστέντα. Αν δεν γίνεται αυτός, θα έχουμε λουλούδια μια ημέρα. Τέλο πάντων, να δημιουργήσουμε πολύ όμορφα λουλούδια που δεν θα κρατούν πολύ. Χρειάζεται αυτού του είδους η συζήτηση. Δηλαδή πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Μακροπεριφερική πολιτική πώς συσχετίζεται με την περιφερική πολιτική και τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. Και μετά στην έκθεση μπορούμε να μπούμε σε λεπτομερέστερη ανάλυση των διαφόρων στατικικών που έχουν προεπιλεγεί για τη ζώνη των Άλπεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Um, ε, αυτή είναι η βασική συζήτηση ε, και το βασικότερο στοιχείο της συζήτησης αυτής είναι οι δικοί σας απόψεις για το πλαίσιο και πώς το βλέπετε για την έκθεσή σας. Και τώρα θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τους πιο εισηγητές και να αρχίσουμε από τον κύριο Γιάκοφσιτς που είναι έτοιμος όπως βλέπω να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να πω το εξή. Την κυρία Μπρέσο την ξέρω επί μία δεκαετία και πλέον και γνωρίζω πολύ καλά το ρόλο της ε, στην περιφέρεια του Πεδεμοντίου, στο Πιεμόντε που ήταν περιφερειάρχης. Ε, είμαι βέβαιος ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ καλά ε, καταρτισμένη, γνωρίζει πολύ καλά την περιφέρειά της η ίδια και τα προβλήματα της περιοχής των Άλπαιων. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω δύο πράγματα τα οποία ανέφερε και ήδη η κυρία Μπρέσο. Πρώτον, η πρωτοβουλία αυτή απορρέει και πηγάζει από τις ίδιες τις περιφέρειες της περιοχής των Άλπαιων. Όπως και η πρωτοβουλία για την Αδριατική και τον Ιόνιο, το Ιόνιο, συγγνώμη, πέλαγος, που από τις ίδιες αυτές τις περιφέρειες γεννήθηκε. Και με εστιάζει στις ανάγκες. Μετά έχουμε τα τρία όχι. Δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχει χρηματοδότηση και δεν υπάρχει νέα νομοθεσία. Τα τρία no στα αγγλικά. Αυτό μπορώ να το δεχτώ να ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι στην πρακτική τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Οι περιφέρειες αυτές που μπορεί να είναι είτε αστικές, ε, είτε κράτη, είτε περιφέρειες, θα δουν και μετά από συνεργασία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλουν να προχωρήσουν και να συνεργαστούν. Και όσοι θέλουν να συνεργαστούν περισσότερο, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται στη δράση τους. Αν θέλουν να δημιουργήσουν περισσότερες δομές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σενετζότο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και καλημέρα σας. Καλώ ήρθατε και από πλευρά η κυρία Μπρέσο που χαιρετίζω το, έργο τη, Εγώ προέρχομαι από το, το, το, Βένετο, στα Ανατολικά, και, ε, από το Πεδεμόντιο η, η Έχει ασχοληθεί με θέματα που τα γνωρίζω και εγώ και οπότε μα είπε τα βασικά ε, θέματα που αφορούν την ε, αλπική περιοχή γιατί αντικειμενικά χρειάζεται να υπάρξει ανάπτυξη όσον αφορά αυτή την ε, απερίμωση. Επομένως ε, χρειάζεται να υπάρξει μία ανάπτυξη η οποία να είναι συμβατή με αυτό που θέλουμε αλλά να μην ξεχνούμε κάποιες βασικές αρχές, βασικούς άξονες. Ε, προέρχομαι από την Βενετία είπαμε οπότε και θεωρούμε για τις Άλπες ότι είναι κάτι σαν ένας τείχος και τα τέχη τη σήμερα ημέρα δεν θα πρέπει να μας εμποδίζουν να πετύχουμε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, να μην εμποδίζουν τη διασύνδεση και θεωρώ ότι σημαντικές στρατηγικές θα πρέπει να υπάρχουν σε σχέση με αυτό το όραμα, να υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που να μπορέσουν να μας βοηθήσουν για αυτούς τους σημαντικούς διαδρόμους, τους ε, θεωρητικούς και τους πραγματικούς. Και αυτές οι στρατηγικές ε, βορρά-νότου ή νότου-βορρά να αφορούν όλη αυτή την περιοχή στα δυτικά που αφορούν το πεδημόνιο και στα ανατολικά που αφορούν το Βένετο. θα πρέπει να ε, ε, είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής αυτής αυτή η διάδρομη. Και επομένως θα πρέπει οι στρατηγικές αυτές να κατατείνουν στο να υπάρξει ανάπτυξη στην ε, περιοχή των Άλπιων. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπε η συγγήτρια, ώστε να μπορέσουμε από κοινού να προχωρήσουμε, να υπάρχει μια συναπόφηση και έτσι τα πράγματα να εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο και να ε, μεταχειριστούμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να υλοποιήσουμε αυτές τις στρατηγικές. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Κύριε Μαρζέ, το λόγο. Ευχαριστώ. Μετά την παρουσίαση και μετά τόσο σαφής αλλά και τόσο λεπτομερής και περιστατωμένη της κυρίας Βρέσο δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Θα ήθελα μόνο να επιμείνω σε ένα σημείο το οποίο και εσείς υπογραμμίσατε και που μου φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι γεγονός ότι η πρώτη σήμερα των Άλπαιων εκάλυπτε ε, ε, μια επικράτεια 190.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και 14 εκατομμύρια κατοίκους. Και τώρα έχουμε ε, διευρύνει αυτή την ε, αντίληψη και έχουμε πάει σε μια μακροπεριφέρεια 450.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 70 εκατομμύρια κατοίκους και όπου συμπεριλαμβάνονται και μεγάλα αστικά κέντρα. Το είπατε και εσείς οι ίδια. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Όχι μόνο για τις ορεινές αλπικές περιφέρειες που θα ευνοηθούν από τις επενδύσεις σε μια κοινή δυναμική και από τις επενδύσεις στις αστικές, δηλαδή των μεγάλων αστικών κέντρων. Και υπάρχει ένας συσχετισμός δυνάμεων εκεί βορρά-νότου στην ε, ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που παίζει το ρόλο του. Ε, μια δεύτερη παρατήρηση, ίσως μια πρόταση που θα μπορούσα να σας κάνω, θα επιθυμούσα να σας κάνω είναι να κάνουμε δεχομένω μία αξιολόγηση των ΕΣΠΑ, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και της τελευταίας προγραμματικής περίοδου, αλλά και της τρέχουσας, έτσι ώστε να εξετάσουμε ε, τα προγράμματα και τις επενδύσεις που γίνονται σε αυτές τις περιφέρειες και να βγάλουμε τα καλύτερα συμπεράσματα έτσι ώστε να χαράξουμε τη στρατηγική μας. Και ένα ακόμα σημείο που είπατε και εσείς η ίδια, σημαντικό για μένα, είναι η διακυβέρνηση. Και εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξισορροπηθεί ο σχετισμός δυνάμεων εκεί στις Άλπες για τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση. Και τέλος η έκθεσή σας θα μπορούσε να επικεντρωθεί και στην εφαρμογή, την υλοποίηση, το είπατε κι εσείς, αλλά και την αξιολόγηση εκ των υστέρων. Και μάλιστα από, την, από το στάδιο της χάραξης και του προγραμματισμού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρκο Τζούλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την συνάδελφο Μπρέσο. Να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι το θεμέλιο αυτή της στρατηγικής οπότε να μπορέσουμε να έχουμε προσθεμένη αξία που αυτό να αφορά τις ε, τοπικές αρχές οπότε θα πρέπει να προσέξουμε τις ε, υποδομές πως από εκεί θα ξεκινήσουμε, πώς θα τις ε, αξιοποιήσουμε, γιατί μιλούμε για περιβάλλον, μιλάμε για ενέργεια που αλληλοσυνδέονται. Οπότε ε, θα πρέπει πρώτα πρώτα να φροντίσουμε ε, την περιοχή και όχι τους πόρους που είναι πεπερασμένοι και όχι το οικονομικό κομμάτι. Οπότε δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την παράδοση κάθε περιοχής. Άρα θα πρέπει να γίνει τέτοια προσέγγιση. Το, το, καινούριο να παντρευτεί με το παλιό ας πούμε. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την διακυβέρνηση και πέραν από τους πόρους θα πρέπει να μην ξεχνούμε το ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές και πρακτικοί. Να λάβουμε υπόψη τις καλύτερες πρακτικές και να προσέξουμε μια τέτοιους προσέγγιση να κάνουμε. Άρα έτσι θα πρέπει από κοινού να προχωρήσουμε. Η πρόεδρος ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα λόγο έχει ο κύριος Μπόγκοβιτς. Είστε σκιώδης συγκητή ή εκ μέρου του. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, έχουμε ακούσει ότι στην Ευρώπη υπάρχουν τέσσερις μακροπεριφέρειες, η Βαλτική και μετά άλλες τρεις. Και μεταξύ αυτών είναι και η περιοχή των Άλπαιων. Εμεί είμαστε μια μικρή χώρα, η Σλοβενία, 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συμμετέχει σε τρεις μακροπεριφέρειες. Και έχουμε λοιπόν κάποια εμπειρία ήδη αποκομίσει, έστω και αν είμαστε μικρή χώρα για, ας πούμε, στην μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου. Έρχομαι τώρα στις Σάλπης και στην έκθεση της κυρίας Μπρέσο. Το Γενάρη ήμουν στο Μπέρτο Μπαϊκράν στη Σλοβενία ε, όπου άρχισε η συζήτηση για την υλοποίηση της ε, σύμβασης αυτής. Συμμετείχα στις εργασίες ε, αυτές Και ήδη στη Σλοβενία οι συμμετέχοντες ήταν από 300 μέχρι 400 από διάφορους τομείς ε, της Παλαιάς Σύμβασης των Άλπαιων. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται πραγματικά προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Ήταν παρούσες και δύο επίτροποι Ευρωπαίες και πολλές πολιτικοί και κυρία Πρέσο ίδια σε αυτή την εκδήλωση και σε αυτή τη διοργάνωση και η συγγήτρια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, στις ορεινές περιοχές. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι η σύμβαση αυτή και η στρατηγική που μας απασχολεί τώρα για τις Άλπεις θα βοηθήσει ε, με πολύ μεγάλη επιτυχία τις περιοχές αυτές που είναι και από τις πιο ανεπτυγμένες στην Ευρώπη. Ο κόσμος θα πρέπει τελικά να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που έχει για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας ε, των ειδών, για τη διατήρηση των υδατίνων πόρων, για την ανάπτυξη της κυκλοφορίας και των συγκοινωνιών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η περιφέρεια των Άλπαιων είναι ε, περιοχή διαμετακόμισης. Ε, επίσης, στη Βόρεια Αδριατική έχουμε λιμάνια που συμμετέχουν και εντάσσονται γεωγραφικά σε αυτή την περιφέρεια. Ο τουρισμός, άλλο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε πόσα πράγματα καλύπτονται Χρειάζεται οπωσδήποτε ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. Είμαστε μια κοινωνία που αλλάζει και θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλες τις προκλήσεις από κοινού. Η ανάπτυξη οικονομική είναι σημαντική, οι διασυνδέσεις, τα είπατε, το περιβάλλον, η ενέργεια. Πάρα πολύ σημαντική στόχη όλοι αυτοί. Και θα πρέπει ο κόσμος επιτόπου να ε, τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά και να τα βλέπει να συμβαίνουν. Είναι πολύ σημαντικό η στρατηγική αυτή να υλοποιηθεί και να αποκτήσει σάρκα και οστά και να γίνει κτήμα των ανθρώπων επιτόπου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε μεγάλε εμπειρίε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το θέμα δεν είναι τι θα κάνουμε εμεί για αυτού του ανθρώπου, αλλά τι θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι 80 με 90 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να επιτυγχάνουν πολλά όταν συνεργάζονται και να υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη, πρόοδος και ευημερία. Με βάση και τη βοήθεια αυτών των στρατηγικών θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Και επομένω να γίνουν πολλά πολύ σημαντικά. Ο κύριος Πανίστερ Ρόι, θέλετε το λόγο. Would you like to take a floor? No. Το λόγο. Just shortly, a couple of remarks. Κάνα δύο σχόλια έχω. Πρώτα, Θέλω να πω ότι πολλά μέρη της περιοχής των Άλπων είναι πολύ πλούσια, πάρα πολύ πλούσια. Η Ελβετία που δεν είναι καν μέλος Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η στρατηγική μας πώς λαμβάνουμε υπόψη την Ελβετία, τη θέση της Ελβετίας. Και άλλες περιοχές είναι πολύ πλούσιες. Ξέρω το Πεδεμόντιο. Είναι ο πλούτος της Ιταλίας εκεί ένα, ένα τμήμα της εργατικής δύναμης, της κινητηρίας δύναμης της Ιταλίας είναι εκεί. Ε. Δεν υπάρχουν μόνο προβλήματα, υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Περί αυτού πρόκειται. Είπατε ότι είναι κάτωθεν προσέγγισης. Όλες οι πολιτικές μας, η περιφερειακή, ε, τον κάτωθεν κινείται. Αφορά την επικουρικότητα. Εδώ εξετάζουμε την δαφική διάσταση. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα και θέλουμε άλλη προσέγγιση. Μιλήσατε για τις διασυνδέσεις βορρά, νότου, ανατολής, δύσης κλπ. Θέλουμε να δούμε τι χρειάζεται. Ο τίτλος της εκθέσεώς σας, κατά την άποψή μου, είναι «Στατηγική Ευρωπαϊκής Ενώσεως» των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. μπορείτε να πείτε ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ενώσης στην όλη προσπάθεια για τη νέα μακροπεριφέρεια. Μπορούμε να μαζέψουμε κάποια μέσα που διατίθενται. Και άλλοι αναφέρθηκαν στη διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να επικρατήσει ούτε η Ευρώπη. Διότι αν επικρατήσει η Ευρώπη τέτοιες μέρες υποστηρίζεται λιγότερο ο λαός χρειάζεται περιορισμένη, πολύ περιορισμένη στρατηγική με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Αν μπορεί να το κατορθώσει αυτό κανείς μέσω μιας προσεγγίσεως διακυβερνήσεως με τα τρία όχι που είχαν διατυπωθεί εκ των προτέρων τότε κάτι τέτοιο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε θετικά αποτελέσματα. Τελευταίο σχόλιο. Στην Επιτροπή την περιφερειακή έχουμε ένα έγγραφο τοποθέτησης όσον αφορά ποια είναι η θέση μας για τις ορεινές περιοχές. Το συζητήσαμε την περασμένη φορά, την τελευταία φορά δεν ήσασταν εκεί και εγώ ρώτησα. Γιατί να μην τα υποβάλουμε στην Ολομέλεια τα διάγραφα, σε μια κοινή συζήτηση. Δεν μπορεί κανείς τον ένα μήνα να αναλύει τις ορεινές περιοχές και ε, την περιοχή των άρμων τον επόμενο μήνα. Ίσως μπορούμε Εκτός να έχουμε γενική και ειδική έκθεση, ίσως πρέπει να συνδέσουμε τις εκθέσεις αυτές ε, όταν πάμε στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε τι τροπή θα πάρουν τα πράγματα. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι διαφορετικές προσεγγίσεις αυτές. Έχουμε πολλά άλλα όρη στην Ευρώπη με εντελώς ε, διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις Άλπεις. Αυτή είναι η προσωπική μου παρατήρηση. Ο κύριος ε, Πόλτσακ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνω στα όσα είπε ο κύριος ε, Μπόκοβιτς και στα όσα είπε ο κύριος Βανίστερλόι, θέλω να πω ότι η περιοχή των Άλπαιων είναι πλούσια, αντιμετωπίζει όμως διάφορα προβλήματα. Είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλες περιοχές στην Ευρώπη. Αναφερθήκαμε στην αστική κινητικότητα και τη σχετική έκθεση που συζητήσαμε κατά παρελθόν. Και σημαντικό μέρος του πληθυσμού ε, μετακινείται και μετεγκαθίσταται. Η περιοχή των Άλπαιων πρέπει να αντιμετωπίσει και την γύρανση του πληθυσμού. Και στην Τσεχία πρέπει να έχουμε παρόμοιο πρόβλημα. Λοιπόν, εξ αυτού έχω κάποιο σχόλιο. Η έκθεση ίσως μπορούσε να εμπνεύσει και άλλες περιοχές, άλλες περιφέρειες που πλήττονται από παρόμοια προβλήματα με άλλες ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με τις Άλπεις. Και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί όχι μόνο από την Επιτροπή μας αλλά και από την Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητεί κάποιος άλλος τον λόγο. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο ονόματα έχω στον κατάλογο. Ανδρέας Μερέιτ της DG Regio και κυρία Φιλομένα Καρβάλιο. Ναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Να πω ότι ευπρόσδεκτη, ευπρόσδεκτα μάλλον τα σχόλια της εισηγήτριας της κυρίας Μπρέσο Μα στήριξε στην όλη προσπάθεια. Να πω καταρχάς ότι βάση της στρατηγικής είναι 7 χώρες. Δύο από αυτές δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσης και έχουμε 48 περιφέρειες. 26 από αυτές είναι της Ελβετίας. Άρα αυτό δημιουργεί επιπλοκές. Έχουμε μια χώρα ΕΟΧ και μια χώρα ΕΖΕΣ. πρέπει να εξετάσουμε και αυτά δηλαδή. Θέλουμε πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για καλύτερο συντονισμό δράσεων και χρηματοδοτήσεων. Δεν είναι μια νέα στιβάδα συνεργασίας, νέο στρώμα συνεργασίας, αλλά είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας, αντιμετωπίσεως προβλημάτων θέλουμε να συμπληρώσουμε τυχόν κενά και όχι να υπάρξει επικάλυψη. Τέσσερα στοιχεία θέλω να αναφέρω. Πρώτον, η στρατηγική εστιάζεται επί αποτελεσμάτων και συγκεκριμένων δράσεων. Δεύτερον, ε, έχει προσανατολισμό προς έργα. Προσανατολίζεται προς έργα. Θέλουμε συγκεκριμένα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν. Τρίτον, θα έχει αποτελέσματα με σωστή ισχυρή ηγεσία. Τέταρτον, εάν δεν διατίθενται οι πόροι συνεχώς και αν δεν διατίθεται προσωπικό, αν δεν διατίθεται χρήματα συνεχώς, αν δεν υπάρχει συνεχής υποστήριξη δεν θα λειτουργήσει γιατί χρηματοδότηση. Υπάρχουν 72 προγράμματα περιφερειακά και εθνικά που στηρίζονται στην περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλοί πόροι μπορούν να κινητοποιηθούν. Θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε τη στατικική με τα μέσα χρηματοδότησης που υπάρχουν. Διακυβέρνηση. Έχει, υπάρχει το πλαίσιο το σωστό. Λεπτομέρειες πρέπει να ρυθμιστούν και να συμφωνηθούν μεταξύ των εταίρων. Σημαντικό στοιχείο σφαιρική προσέγγιση. Προτείνουμε μια βάση που να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Να εκπροσωπείται η κοινωνία των πολιτών και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Να εκφράζονται. Τέλος. Τι επιδιώκουμε. Να λειτουργήσει άμεσα στρατηγική. Ποια είναι τα καλά νέα. Οι ομάδες δράσης που θα κινούνται επιτοπίως με τους εμπειρογνώμονες έχουν ήδη συσταθεί. Πανέτοιμες είναι για να εφαρμόσουν τη στρατηγική και τις δράσεις που συμπεριλαμβάνουν το σχέδιο δράσης. Αυτά είναι τα καλά νέα. Και βλέπουμε ότι αυτή η στρατηγική ε, μας δίνει κάποιες υποσχέσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρεσό, θέλετε να απαντήσετε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, λέει η κυρία Μπρέσο, για τις θετικές τους παρατηρήσεις και για όλες αυτές τις προτάσεις τους που διατύπωσαν. Σίγουρα πρόκειται για ένα ζήτημα που ανέκαθεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η άλπιση είναι πέρασμα ιστορικού χαρακτήρα στην Ευρώπη. Ε, πάρα πολλά πρέπει να γίνουν και πάρα πολλά να ολοκληρωθούν όσα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Οπότε αυτό είναι ένα πραγματικό στοιχείο της ε, στρατηγικής ότι δηλαδή θα πρέπει να ληφθούν κάποιες ε, αποφάσεις και οπότε θα πρέπει και οι σχετικές αποφάσεις να υλοποιηθούν. Οπότε η στρατηγική θα πρέπει να λάβει υπόψη τους μεγάλους άξονες του Ανατολής Δύσης. Όλα αυτά θα ωφελήσουν τις περιοχές, τις ε, κοντινές των Άλπαιων και τις ε, περιοχές που βρίσκονται στις Άλπες και επομένως κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Πρόκειται για άξονες επίση μεταφοράς, αλλά όχι μόνο γιατί είναι και θέμα ηλεκτρική ενέργεια, πρόκειται για αυτά τα εφή δίκτυα που υπάρχουν και θα πρέπει να καλυφθούν επομένω οι αλπικές περιοχές που θα μπορούσαν όχι μόνο να καταναλώνουν αλλά και να παράξουν ενέργεια και επίση αυτό έχει σχέση και με το, το διαδίκτυο που θα πρέπει και εκεί να στηθεί ε, αλλιώς η αγορά θα καταρρεύσει γιατί χωρίς να, να υπάρξει κάποιο είδου κρατική παρέμβαση δεν γίνεται να προχωρήσουμε. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να ελεγχθεί αν γίνεται και επομένως είναι θέμα σύνδεσης ή διασύνδεσης και έτσι να έχουμε μεγάλες επενδύσεις που να καλύψουν το σύνολο της αλπικής περιοχής. Αυτές οι συνδέσεις, διασυνδέσεις που αποφέρουν αποτελέσματα ε, και για τις σχετικές περιοχές και μόνο για το σύνολο της ε, Ένωσης. Επομένω, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, όπως εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν, ότι τώρα εξεργάζεται την στρατηγική αυτή κάτι άλλο τώρα το οποίο φύγει από τους συναδέλφους είναι το εξής. Η σχέση μεταξύ τις ορεινές περιοχές και τις παιδινές. Και πολύ σωστά να καλύπτονται και η ΜΕΝ και η δε από τη σχετική στρατηγική. Πολύ σημαντικά γιατί πρόκειται για κάποια πρόκληση, για το πρόβλημα δηλαδή του πώς θα υπάρχει εξισορρόπηση των αναγκών βορανότου, να ληφθούν υπόψη επομένως αυτές οι ορεινές περιοχές οι οποίες ε, έχουν μια μεγάλη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και που να μην αδικηθούν σε σχέση με τις παιδινές περιοχές. Να υπάρξει προστασία Πάντοτε επομένω ζούσε ο κόσμο στι άλπε, πάντοτε διέσχισε τι άλπε. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει για να ε, αξιοποιήσουμε αυτό το εγχείρημα. Επίση να δούμε και τι γίνεται και με την αλλαγή του κλίματο. Μια που υπάρχουν τώρα πολύ σημαντικά προβλήματα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος έχει αρχίσει να σπανίζει το χιόνι στις Άλπες. Άρα θα πρέπει να δούμε, ε, να προβληματιστούμε τι είδους ε, πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης θα έχουμε στις ε, Άλπες. Πάρα πολλά άλλα θέματα αναφέρεται από τους συναδέλφους πάνω στα οποία θα πρέπει να συνεργαστούμε και πρώτα όλα γιατί θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική για την περιοχή των Άλπαιων και όχι για όλα τα βουνά γιατί υπάρχει ιδιοτυπία αυτή τη περιοχή. ή τέλο πάντων κάθε βουνό έχει τι δικέ του ιδιορυθμίε. Υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετική ιστορία. Άλλα χαρακτηριστικά στα Πυρηνία και άλλα στα Καρπάθια. Άρα και θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια στρατηγική από τη βάση προς την κορυφή και οπότε επίσης υπάρχει και μια προϊστορία συνεργασίας για τέτοιες πολιτικές. Άρα θα πρέπει αυτό να το ενισχύσουμε, να το υποστηρίξουμε και να έχουμε ένα εργαλείο το οποίο το έχει εξατομικεύσει η Ένωση. Οπότε, στα πλαίσια της στρατηγικής έχουμε εδώ εμπλεκόμενες δύο μη ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος πάντων, που δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίχτενστάιν και Ελβετία είναι χώρες του ΕΟΧ, ανήκουν στο Σέγγεν και έχουν μία μακρά παράδοση συνεργασίας και πρόκειται για κάποιες ε, μακροπεριφερειακές πολιτικές και στρατηγικές. Οπότε εδώ θα πρέπει να εμπλακούν αυτές οι χώρες. Οι χώρες οι οποίες δεν γίνεται να απουσιάσουν από τη στρατηγική για τις άλλες. Είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτής για αυτή τη στρατηγική, άσχετα από τις άλλες μακροπεριφερειακές στρατηγικές, έχει άλλα χαρακτηριστικά η Παιδιάδα και άλλα το βουνό. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το ατού της μακροπεριφερειακής στρατηγικής, ότι ξεκινά λαμβάνοντας υπόψη ε, την ταυτότητα. Είναι κάτι το οποίο προϋπάρχει πριν χαραχτεί αυτή η στρατηγική. Άρα ξεκινάμε εδώ την συνεργασία και λέμε για περιφερειακή συνοχή, αυτό το οποίο έχει ενσωματωθεί στην συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά δεν έχουν δοθεί ξεκάθαροι ορισμοί. Κατά τη γνώμη μου όμως αυτές οι στρατηγικές, οι μακροπεριφερειακές, αποτελούν ε, έναν ορισμό, μια συγκεκριμενοποίηση του τι είπα να πει ε, εδαφική συνοχή στην Ευρώπη. Αν θέλουμε η Ευρώπη να συνεργάζεται, να το δούμε αυτό, ενισχύει γιατί έχουμε τώρα κάποιο είδους μαντάτα, μάλλον ε, μελανά. Τέλο πάντων, θα πρέπει να μην τα ξεχάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, εάν πραγματικά θέλουμε να υπάρξει συνεργασία. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδων χιλιόμετρων που καλύπτονται από τις ε, περιοχές αυτές. Βέβαια, έχουμε βέβαια και κάποια πιο δύσκολα στοιχεία όπως την απερίμωση, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα προσβασιμότητας κάποιες υπηρεσίες, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε διάλογο μεταξύ ε, των ε, μεγάλων πόλεων της Παιδιάδας και των πιο ορεινών περιοχών. Γιατί βέβαια οι μεν ε, βοηθούν τους δε. Ο τουρισμός ας πούμε και άλλοι πόροι που στέλνει ούτως είπε ο μεν στον ΔΕΑ, δηλαδή η παιδιάδα στο βουνό. Αλλά να δούμε και το θέμα του τουρισμού σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή ε, διαχείριση, ισχυρή πρωτοπορία. Είδαμε τι έγινε στην ε, Σλοβενία χωρίς ε, κάποιο είδου ισχυρή διακυβέρνηση δεν μπορούμε να συνδυάσουμε τους ε, σχετικούς πόρους. Όχι μόνο τους οικονομικούς, αλλά και ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Να, είδαμε τι ισχύει σε αυτό το πανεπιστημιακό δίκτυο για τη σχετική στρατηγική. Άρα θα πρέπει να υπάρξει σχόλιο και πανεπιστημιακή αυτών των μετόπων όπως η αλλαγή του κλίματος, τι γίνεται με τις βιώσιμες οικονομίες, πολύ σημαντικά αυτά για τις ορεινές περιοχές. Εδώ δεν λέμε για μια περιοχή της Άλπης που είναι καθυστερημένη. Υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι που ξεπηδάνε από τις Άλπεις... άρα Υπάρχει το θέμα εδώ της καινοτομίας, όπως και το θέμα της διατήρησης της παράδοσης. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν, πρέπει να υπάρξει συνεργασία για την αλπική περιοχή και να υπάρξουν συγκεκριμένα σχέδια ή προγράμματα και προς τα εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούν οι οικονομικοί πόροι οι οποίοι χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν με ευθεία και με πνεύμα συνεργασία. Αυτό είναι βέβαια το, πιο δύσκολο γιατί πρόκειται για περιοχή πάρα πολύ εκτεταμένη. Οπότε χρειάζεται κανείς να έχει αφοσίωση και να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για τη συνεργασία. Εμείς το τονίζουμε. Βέβαια, για να υπάρξει στιβαρή ηγεσία σε αυτήν την πολιτική διακυβέρνηση, θα πρέπει αυτή η διακυβέρνηση να λαμβάνει υπόψη το ότι θα πρέπει να ε, δοθεί ιδέουσα σημασία στις ε, περιοχές αυτές που ενδιαφέρονται γιατί μιλάμε για πάρα πολύ ε, μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαμε τους υπουργούς αυτών των χωρών που δεν δίνανε το, τη, τη σχετική σημασία. Όμως οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις αυτών των περιοχών, όλοι οι εμπλεκόμενοι με την ευρεία σημασία ενδιαφέρονται. Σωστό. Άρα χρειάζεται μια διακυβέρνηση πάρα πολύ στιβαρή, ούτως ώστε όλα να λειτουργήσουν σωστά. Πάλι σας ευχαριστώ για αυτή την έκθεση που θεωρούμε ότι θα κινητοποιήσει τα πράγματα, αλλά θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε και να δούμε τι κατεύθυνση θα πάρει αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση αυτή. Και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα μας, στη μέρη σε διάταξη. Το Σεπτέμβριο του 2015 η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα με Ατόπο με Αναπηρία ενέκρινε μια έκθεση και σχετικά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής της σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ. Έγινε διάλογος Ηνωμένων Εθνών Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνέχεια για μια σειρά θεμάτων που κατήρθησε η αρμόδια επιτροπή και η δική μας επιτροπή απασχόλησης μαζί με τη ΛΥΜΠΕ και την ΠΕΤΗ και τώρα γίνεται έκθεση για την κατάσταση των πραγμάτων ε, της εφαρμογής ε, της σύμβασης αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, η είναι η κυρία Χέτ, συντάκτερης συντάκτρια της νομοδότησης, δυστυχώς ε, κολλείεται σήμερα και απουσιάζει, οπότε θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κρέλ που θα παρουσιάσει το σχέδιο ε, γνωμοδότησης της κυρίας Χέντ εξ ονόματός της. Προτείνω προθεσμία για τις τροπολογίες 22 ε, του μηνός Φεβρουαρίου, επόμενη Δευτέρα το μεσημέρι για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε το Μάρτιο την έκθεση, τη γνωμοδότηση στη δική μα Επιτροπή. Έχουμε χρονικό περιορισμό δυστυχώς ε, και δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Κρέλ και μετά στους εκπροσώπους και τους σχεδόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Λυπάμαι πάρα πολύ που η κυρία Χέτ σήμερα και απουσιάζει και εγώ προσωπικά πριν από μια μισή ώρα το έμαθα όταν έφτασα στις Βρυξέλλες, δηλαδή δεν είμαι και ιδιαίτερα προετοιμασμένη και πραγματικά διαβάζω αυτά που μου έγραψε η κυρία Χέτ και τίποτα άλλο. Πιστεύω όμως ότι δεν είναι τόσο περίπλοκο το θέμα διότι στους κανονισμούς για τα ταμεία. Τα τελευταία χρόνια κάναμε πολύ καλή δουλειά και προσέξαμε πάρα πολύ. Φροντίσαμε πάντα τους ανθρώπους με αναπηρία. Με ιδιαίτερη πάντα προσοχή και επιμέλεια. Τα έχουμε εντάξει στην νομοθεσία και της πολιτική συνοχή στην Ευρώπη. Θα τα διαβάσω τώρα αγγλικά για να μην τα μεταφράζω τώρα έτσι δύο φορές γερμανικά και τα λοιπά, για να σας πω τι είπε η κυρία ε, Χέτ. Η δική της φιλοδοξία ήταν να επικεντρωθεί στα σημαντικότερα ζητήματα από τη δική μας κοπιά της περιφερειακής πολιτικής. Τονίζει στην γνωμοδότησή της η κυρία Χέπ ότι ο κοινός κανονισμός έχει άρθρα όπως το 7 και το 96-7 που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες, τη μη διάκριση και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες παντού στην εφαρμογή και την υλοποίηση ε, των κονδυλίων από τα επενδυτικά και τα διαστατικά ταμεία. Στα γενικά προγράμματα και στα ΕΣΠΑ ειδικότερα. Αυτά τα άρθρα είναι σημαντικά και θα πρέπει να διέπουν ε, τη χρηματοδότηση. Δεύτερον, η γνωμοδότηση καλεί τα κράτη-μέλη αλλά και τις περιφέρειες και τις ΟΤΑ να αυξήσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της πρόληψης των διακρίσεων και του αποκλεισμού ατόμων με αναπηρίες από διάφορους τομείς και θα πρέπει να προάγεται και ίση ε, πρόσβαση στην υγεία. Ένα σημαντικό στοιχείο στην γνωμοδότηση έχει να κάνει με τις παρατηρήσεις που έκανε η αντίστοιχη επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Καλή η γνωμοδότηση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο για τους τομείς αυτούς και όπως αυτοί αναφέρονται ε, στην αρχική έκθεση. Και τέλος, η γνωμοδότηση τονίζει επίσης ότι η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθούν ε, οι επενδύσεις ε, υποδομή ε, για να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο και το επίπεδο ζωής των ανθρώπων αυτών. Επίσης μας ανησυχεί η ιδρυματοποίηση και οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών σε ιδρύματα. Και λέει η κυρία Χέτ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία στη γνωμοδότηση και περιμένει με χαρά να τη συζητήσει με τους και ηγητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθούν οι σκιώδεις συζητητές. Ο κύριος Πόλτσακ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι αρκετά σύντομη και περιεκτική, αλλά είμαι πεπισμένος ότι ανταποκρίνεται πολύ καλά στα όσα αναμενόταν και αναφέρει σωστά όλα τα ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή δεν απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή στρατηγική για ε, τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το να διέπεται σε κοινοτικό επίπεδο το πρόβλημα αυτό. Τα άτομα με αναπηρία κατά το παρελθόν μπόρεσαν να ευνοηθούν από την επιτευχθήσα πρόοδο κατά την περίοδο αυτή. Στην έκθεση αναφέρεται ότι ένα άτομο στα έξι στην Ευρώπη έχει κάποιο πρόβλημα, κάποια αναπηρία, αρκετά σημαντικό ποσοστό Υπάρχουν διάφορα επίπεδα αναπηρίας, λίγο πολύ σοβαρά, αφορά περίπου 80 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή, στην οικονομική ζωή, λόγω κάποιων εμποδίων που αντιμετωπίζουν και που μπορεί να τους οδηγήσουν και μέχρι στη φτώχεια. Το μέσο εισόδημα αυτών των ανθρώπων ε, είναι περίπου στο 70% του, υπολείπου, του εισοδήματος του υπολείπου πληθυσμού. Και αυτό δημιουργεί, ε, διότι έχουν και προβλήματα όσον αφορά τις αμοιβόμενε εργασίες. Και πολλά από αυτά τα άτομα πάνω από 50, που είναι πάνω από 50 ετών ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα που παρεμποδίζουν τη δραστηριότητά τους και πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν ε, πολύ σημαντικό βαθμό αναπηρίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη γύρανση του πληθυσμού, ε, πιστεύω ότι θα αυξάνεται ο αριθμός αυτών των ανθρώπων. Αυτά παρουσιάζει το έγγραφο ε, και η έκθεση της ηγήτριας και βλέπουμε σε ποιο βαθμό αυτό το θέμα είναι σημαντικό λόγω των τάσεων που υπάρχουν. Και λόγω των τάσεων θα αυξάνεται η σημασία του κειμένου και θα δείχνει σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις της πολιτικής συνοχής μπορούν να παίξουν όλο και σημαντικότερο ρόλο. Να συμπιστήσω την προσοχή και επί του εξή. Στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική βοηθείας που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία, ζητάμε ε, να υπάρξει αποθεσματοποίηση των, της περίθαλψης που παρέχεται και στα πλαίσια ενός εγγράφου που υθετήθηκε από το Κοινοβούλιο πέρσι ε, επί του θέματος των διαφόρων περιθεριοποιημένων κοινοτήτων ακολουθείται παρόμοια προσέγγιση. Εκείνο το έγγραφο απευθύνεται κυρίως στα κράτη-μέλη. Ίσως να υπάρχει και πρόβλημα συντονισμού των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ενώσης στον τομέα. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμός, πιο ανοιχτή προσέγγιση και χρειάζεται εμβάθυνση της ανάλυσης. Κυρία εισηγήτρια συνέταξε μια έκθεση σύντομη, περιεκτική, πληρέστατη και προσωπικά. Θα υποβάλω μία ή δύο τροποποίησεις να υποβάλω, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή βάση για συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η δυο τροποποιησεις να υποβαλω αλλα πιστευω οτι ειναι παρα πολυ καλη βαση για συζητηση ευχαριστω πολυ λεει προεδρος Ναι, γνωρίζω. Στην κυρία Ρέντκε και στον κύριο Μάτο θα δώσω το λόγο. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Στην κυρία Νταμάτο μετά, συγγνώμη. Συγγνώμη, ξεπλάγιν γιατί προχωρήσαν πολύ γρήγορα. Έλεγα ότι θα υπάρξουν και άλλοι σκιώδεις το μιλούσαν. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, γνωμοδότηση αυτή. Είναι πολύ καλή αφετηρία, διότι όπως προαναφέρθηκε, το θέμα της εντάξεως των ανθρώπων με αναπηρία θα πρέπει να φωτίζεται περισσότερο, διότι μπορεί να ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά στην υλοποίηση συμβάσεως του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και σχετικά με την πράξη της προσωσιμότητας για τη στρατηγική για την οριζόντια ισότητα. Χρειάζονται κοινέ προσπάθειες για να προχωρήσουμε και να μπορούμε να συμπεριλαμβάνουμε τα άτομα με ε, αναπηρίες σε όλες τις πτυχές κοινωνίας μας. Και όλα αυτά τα μέτρα μπορούν πράγματι να έχουν οικονομικές συνέπειες το βλέπουμε από την οπτική γωνία της Ρέτζιο, δηλαδή πώς να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να ελοπίσουμε τους στόχους. Είναι σημαντικό το έγγραφο. Όπως είπα, είναι μια πολύ καλή αφετηρία. Σε κάποια σημεία μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις. Θα θέλαμε να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες ή παραδείγματι. Να προσέξουμε όλος ιδιαίτερος οι πόροι Ευρωπαϊκής Ενώσεως να μην χρησιμοποιούν σε, για ε, μέτρα που οδηγούν σε απομόνωση. Τα κάτι μέρη που χρησιμοποιούν πόρου τη Ευρωπαϊκή Ενώση με έναν τρόπο που ίσω να αποκλεί ανθρώπου με αναπηρία, ε, να ξεκινούμε και διαδικασίε κατά παράβαση για να υπάρχει σωστή χρήση ε, των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, σημαντικό το σημείο που αναφέρεται ήδη στο σχέδιο γνωμοδοτήσεω. Αλλά πρέπει να τονιστεί. ισότητα και η μη διάκριση είναι βασικέ αρχέ και οι πόλεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως καταπολεμούν τη διάκριση, κυρίως στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην περίθαψη υπηρεσίες υγείας και σε όλα τα στάδια της χρήσης των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άνθρωποι με αναπηρίε και στη λήψη αποφάσεων. Διότι οι άνθρωποι με αναπηρία είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα, που πρέπει να επιφέρει αλλαγές η κοινωνία για να μπορούν να εντάσσονται καλύτερα. Τέλο, Ίσως χρειάζεται μια συμπλήρωση, μια προσθήκη. Σε τοπικό επίπεδο χρειάζεται πιο ανοιχτή προσέγγιση όσον αφορά τις υπηρεσίες, να συμπεριλαμβάνονται οι άνθρωποι με αναπηρία, να απολαμβάνουν πλήρως των δικαιωμάτων τους ε, σαν πολίτες της Ευρωπαϊκής Προσβλέπω στις συζητήσεις με συναδέλφους ε, και κυρίως στις συζητήσεις με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταμάτο και μετά ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια. Την συντονίστρια για τους σοσιαλιστές. Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως γνωρίζουμε. Έχει προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε αυτή τη την για τον Δεκέμβριο του 2010. Πρόκειται για τα άτομα με αναπηρία. Βλέπουμε ότι είναι πρωτόκολλο αυτό το πλέγμα προστασίας και, και υπεγράφει αυτό το πρωτόκολλο, αλλά πρέπει και να επικυρωθεί. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι πρωτοβουλίες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα άτομα ειδικέ ανάγκες. Οπότε θα υπάρχει εδώ πέρα θέμα ε, περιφερειακό, θέμα οικονομικό και κοινωνικό για τους Ευρωπαίους αυτούς οι οποίοι πάσχουν κάποια αναπηρία. Ακριβώς όμως έχουμε κάποιες περικοπές χωρίς προηγούμενο λόγω της κρίσης. Περικοπές και στην κοινωνική πρόηνα. Οπότε οι ανάπηροι τώρα βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής ε, περιθωριοποίησης και φτώχειας. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα τους δώσουμε μια ανεξαρτησία στην ε, ζωή τους, μια θέση στην ε, κοινωνία. Όλα τα υπόλοιπα τα προβλέπει η σύμβαση του ΟΗΕ. Υπάρχουν επίσης μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτήν την ε, σύμβαση του ΟΗΕ για τους αναπήρους. Εν κατακλείδη νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επικυρώσει ε, αυτό το πρωτόκολλο. Αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία δεν το έχουν πράξει ακόμα. Επίσης υπάρχει και ένα προαιρετικό πρωτόκολλο που επισυνάπτεται σε αυτήν την ε, σύμβαση του ΟΗΕ που είναι σημαντικό γιατί έτσι η, η Επιτροπή CPRD του ΟΗΕ ε, θα μπορούσε να έχει αρκετούς πόρους για ομάδες και για εξατομικευμένες περιπτώσεις να τους βοηθήσει και έτσι να υλοποιηθεί αυτή η σύμβαση. Και να έχουμε αυτή την οργάνωση φωτοφορία European Disability Forum. Οπότε το νωρίτερο δυνατόν θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες με την προσυπογραφή και επικύρωση αυτού του ε, πρωτοκόλλου. Κύριος σας ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος και εγώ του κυρίου Τάκουλα που είναι ο δικός μας και ο θα ήθελα να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας. 18 εκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζεται ότι είναι άτομα με ειδικέ ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άνθρωποι με αναπηρίες. Αυτό τι δείχνει. Πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόζουμε την ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες. Παντού, σε όλα τα κράτη-μέλη, με τρόπο αποτελεσματικό. Αυτό επίσης σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, πρέπει να αλλάξουμε εκπαίδευση, πρέπει να αλλάξουμε παιδεία, πρέπει να αλλάξουμε ε, μυαλά. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχουν φραγμοί όχι μόνο στα μυαλά αλλά και στην πράξη. Ε, φυσικά εμπόδια. Φυσικά και τα εμπόδια τα νόητα είναι σημαντικά, αλλά επίσης σημαντικά είναι και τα φυσικά αντικειμενικά που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα. Έχουν γίνει ήδη πολλά, αλλά παραμένουν τα εμπόδια πολλά. Είμαστε απόλυτοι. Ε, ζητούμε να εφαρμόζονται ε, αυτά παντού σε όλα τα κράτη-μέλη για να ε, υπάρξει και η απαραίτητη δράση και χρηματοδότηση. Βέβαια η χρηματοδότηση είναι πρόβλημα. Για την άρση των φυσικών εμποδίων δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από τη χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, που έχουν αναπηρία. Το είπα από την αρχή. Είναι πάρα πολλοί οι πολίτες. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει να λάβει το λόγο, αλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Γκρέιντς, σωστά το είπα. Ευχαριστώ. Γκρέιντς το όνομά μου. Γαλλικότατο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σημειώνω εν ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μεγάλη ικανοποίηση την υποστήριξη των διαφόρων που πήραν τον λόγο στην Επιτροπή σας. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα θέμα σημαντικότατο για μας. Είμαι επικεφαλής μονάδας ματάρχης που ασχολείται με την ε, πολιτική και τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία στην Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση. Επανερχόμενοι στο θέμα τώρα. Ασχολούμεθα πολύ με την πολιτική αυτή και την προάσπιση των ανθρώπων με αναπηρία. Και για μας είναι σαφές ότι οι πτυχές που υπερασπίζεστε στην περιφερική πολιτική είναι πολύ σημαντικές για να προχωρήσουμε στο έργο μας. Όλα αυτά που είπατε μας δίνουν τη στήριξη που χρειαζόμαστε για την χρήση των ιδιωτικών ταμείων και των ευρωπαϊκών επενδύσεων που υπάρχει μια ρήτρα ρεσιμότητα στη χρήση αυτών. Έχει αρχίσει η εφαρμογή του νέου προγραμματισμού 2014-2020, αλλά βλέπουμε μία ευαισθητοποίηση των κρατών μελών στα προγράμματα που υποβάλλουν για αυτό το θέμα. Και γίνονται πιο συγκεκριμένα πράγματα. Μιλώ τώρα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όσον αφορά το ΦΕΝΤΕΡ, παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο τη εξέλιξη εκεί. Όταν μιλάμε για αποθεσματοποίηση, αποθεσμοποίηση μάλλον, χρειαζόμαστε δομές και υπηρεσίες. Όλα όσα στηρίζουν στην εφαρμογή της συμβάσεως είναι καλά. Σημειώνουμε όλα όσα υπόθηκαν εξ προθέσει υποβολή τροπολογιών σωστά τα σχόλια όσον αφορά την κύρωση του πρωτοκόλλου Είναι περίπλοκο ζήτημα. Συζητείται ακόμα. Ε, υπάρχουν νομικές πτυχές που συζητούνται. Εδώ δεν μπορώ να σας δώσω πληροφορίες. Η συζήτηση είναι αρκετά εν, εντατική μάλλον που διεξάγεται. Τι άλλο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ελπίζω να κάλυψα λίγο πολύ τα πάντα. Είπαμε η αποδρυματοποίηση είναι κάτι που πιστεύω ότι η κυρία Στίβενς, η συγγήτρια, θα το τονίσει ιδιαίτερος. Είναι σημαντικό για μας, για την Επιτροπή Απασχόλησης επίσης. Αυτά. Συγγνώμη που τα είπα συγκεχημένα αλλά έφτασα από το Συμβούλιο που γινόταν και συζητήσεις εκεί, βλέπετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που έκανα λάθος με το όνομα. Για μία ακόμη φορά ζητώ συγγνώμη. Ο κ. Βαν Νίστελ Ρόι θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Ε, ε, δίσταζα γιατί ε, οι κάτω χώρες δεν έχουν κυρώσει αυτή τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία. Τώρα αυτό το καιρό το συζητούμε. Και θα είχε νόημα να δούμε πώς έχει διατύπωση το σημείο 6 στη γνωμοδότησή μας ε, όπου λέμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κονδύλια ε, ευρωπαϊκά για την αποϊδρυματοποίηση και ε, τις υπηρεσίες. Σωστό είναι αυτό, αλλά μήπως να εξηγήσουμε ποια είναι τα κονδύλια αυτά που έχουμε υπόψη μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κυρίως. Και θα πρέπει να το πούμε αν εννοούμε αυτό. Και πολλά από τα πράγματα αυτά είναι στα χέρια των κρατών μελών που ασκούν την κοινωνική πολιτική. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Δεν ξέρω, μήπως να το κοιτάξουμε και αυτό και να φροντίσουμε να το πούμε πιο συγκεκριμένα, να μην ε, φουσκώσουμε πάρα πολύ τις προσδοκίες γιατί η αποϊδρυματοποίηση είναι μια διαδικασία που διεξάγεται παντού στην Ευρώπη, ε, όπου υπάρχουν πολλά ιδρύματα ε, με άτομα με αναπηρία που σιγά σιγά φεύγουμε από αυτή την προσέγγιση και αποκεντρωνόμαστε. Και οι πολιτικές αυτές εν μέρη είναι δική μας αρμοδιότητα, όχι ο απολύτως. Δεν ξέρω μήπως να το δούμε ξανά το κείμενο. Η Πρόεδρος, ναι, είμαι βέβαια ότι θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε και τροπολογία εσείς ε, μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου την άλλη Δευτέρα όπως είπαμε που λύγει η προθεσμία. Η κυρία Κρέλ, έχετε το λόγο. Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ε, εντατική σας συμμετοχή και τη δραστήρια θα τα διαβιβάσω στην κυρία Χέτ για το τελευταίο σχόλιο του Λάμπερτ Βανίστερ Ρόι. Νομίζω στην παράγραφο 1 και την αναφορά που γίνεται στο άρθρο 7 και στο 96 είναι ξεκάθαρο για το ποιο τομεί ε, αφορά και ενδιαφέρεται. Είναι γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Δεν θα μπούμε στα χωράφια της κοινωνικής πολιτικής των κρατών μελών. Οπωσδήποτε θα πρέπει να συνεισφέρουν εκείνοι περισσότερο αλίμονο για ε, τους ανθρώπους με αναπηρίες. Εμείς μιλούμε στα πλαίσια μόνο των δικών μας αρμοδιοτήτων με τα διορθωτικά ταμεία. Πάντως έχετε όλη τη δυνατότητα, κάνετε και τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος και τώρα ε, πρέπει να σας πω ότι τελείωσε αυτό το θέμα και πάμε στο επόμενο. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκνε μια κατεξοδότηση πράξη ε, με βάση την πέμπτη υποπαράγραφο του άρθρου 122.2 ε, του κοινού κανονισμού για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάποια ποσά που θα πρέπει να ανακτηθούν από τα κράτη-μέλη σύμφωνα με το άρθρο 122 και με βάση ποια παράγραφο γίνεται αυτό για τα μη ανακτήσιμα ποσά. Σε όλες τις γλώσσες το έλαβε το Κοινοβούλιο στις 29 Ιανουαρίου και σας διαβιβάστηκε από τη Γραμματεία με mail την 1η του μηνός Φεβρουαρίου. Θα ήθελα να σας θυμίσω τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί. Το Κοινοβούλιο μπορεί να προβάλλει αντίρρηση εντός διμήνου ε, από την ημερομηνία κοινοποίηση της κατεξοδότηση πράξης. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να εγκρίνει ψήφισμα που θα έχει υποβάλει αρμόδια επιτροπή και θα αθορίζει τους λόγους ε, για τους οποίους έχει αντίρρηση. Αυτά είναι όλα στο άρθρο 105. Εάν επιθυμεί η Επιτροπή μας μπορεί να ζητήσει παράταση της ε, περίοδου αυτής του διμήνου, εάν δεν αναλάβουμε καμία δράση, θα θεωρηθεί εγκεκριμένη η κατεξοδότηση πράξη μετά την παρέλευση του διμήνου. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Dirk Πέτερς από τη Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο για να μας εξηγήσει σύντομα το πεδίο εφαρμογής και ε, τον σκοπό της κατεξοδότηση πράξης και μετά θα αποφασίσουμε για το τι μέλη γενέστε. Το λόγο έχει ο κύριος Πέτερς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο στόχο τη και της ουδέτης πράξης είναι να καθοριστεί κατά πόσο αυτά τα μήνα κτίσιμα ποσά θα πρέπει να καλυφθούν από τα κράτη-μέλη ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επανειλημμένα τα έχουμε στήσει αυτά με των κρατών μελών και το θέμα είναι πως κρατημέλη σε πρώτη φάση είναι γίνα αρμόδια ώστε να μπορέσουν να διορθώσουν ή και να προλάβουν ή και να καλύψουν ε, αυτή την υπόθεση ε, των παρατυπιών και να καλύψουν αυτά τα ανακτήσιμα πόσα εάν σχετικές διαδικασίες δεν πιάσουν τόπο τότε είναι δυνατόν να ζητηθεί αυτά τα ποσά να καλυφθούν από τον προπολισμό της Ένωσης εκτός εάν ε, υπάρχει βαρία ή ελαφρά αμέλεια ή απλό λάθος. Οπότε υπάρχει μια σχετική διαδικασία η οποία προβλέπεται για το πώς θα γίνει αυτό. Και εάν δεν κάνει τίποτα μέχρι κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τότε καλύπτεται ε, το σχετικό ποσό από τον και η κατεξοδότηση πράξη ορίζει ποια είναι τα κριτήρια τα οποία ορίζουν ε, το κατά πόσον το κράτος ε, μέλος έχει ενεργήσει με την δέουσα επιμέλεια. Όταν πληρούνται αυτή η προϋπόθεση, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πιστοποιεί ότι όντως ενήργησε επιμελώς το κράτος μέλος. Έχουμε και το σχέδιο κειμένου νομοθετικής πράξης που προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη διηγούνται να αποφασίσουν ότι δεν θα ανακτήσουν αυτά τα ποσά εάν μιλούμε για ποσά κάτω των 250 ευρώ σε περίπτωση προγραμμάτων συνεργασίας οπότε τα κράτη-μέλη έχουν συμμετάσχει σε αυτό το πράγμα μπορεί να αποφασίσουν ότι δεν θα προβούν στην ανακρίση των σχετικών ποσών. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Κύριε συνάδελφοι, θέλετε το λόγο. Ο κύριος Φανίστελ, Μάλιστα. Θα λάβουμε υπόψη αυτή την ενημέρωση γιατί Φαντάζομαι είναι σημαντικό να γίνει συζήτηση εις τους συντονιστάς. Οπότε και θα πρέπει να προβληματιστούμε και να συνεργαστούμε με τους ε, συνεργάτες με την Γραμματεία της Επιτροπής και να επανέλθουμε. Καλώς λέει Πρόεδρος. Θέλει άλλο το λόγο. Όχι. προτείνω στην Επιτροπή να μην ζητηθεί παράταση Αυτή τη προθεσμίας της δίμηνη για υποβολή ένσταση. Και Τρίτη, 20 Δευτέρου να είναι η κατακλητική ημερομηνία το μεσημέρι. Ούτω ώστε οι συνάδελφοι να στείλουν τις ε, ενδεχόμενε ενστάσει του για αυτή την ε, πράξη. Συμφωνείτε, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα κάνουμε. Επομένω αυτό και θα κάνουμε όσον αφορά αυτού του είδου τον κατεξοδότηση κανονισμό, κατεξοδότηση πράξη. Δεν θα ζητηθεί παράταση και θα ισχύσει αυτή η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ενστάσεων. Και τώρα. Mm. Πέρασε της ε, ανοιχτής συνεδρίασης. Παρακαλώ όλοι εκείνοι που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στη συνεδρία των συντονιστών να εγκαταλείψουν την ε, αίθουσα. Και θα συνεχίσουμε με την συνεδρίαση των συντονιστών. Thank you.